Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf die heutige Sitzung des Haushaltskontrollausschusses eröffnen. Es ist die erste Sitzung unseres Ausschusses im neuen Jahr. Σας καλωσορίζω, σας εύχομαι καλή χρονιά σε όλους και σας και στην οικογένειά σας με υγεία, ειρήνη και επιτυχίες στο νέο έτος. Εύχομαι και στην Επιτροπή μας ε, και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιτυχία στο δύσκολο έργο μας ε, ζούμε εποχές ε, δημοσιονομικών κρίσεων στα κράτη-μέλη και έχουμε πολλή δουλειά εδώ στην Επιτροπή με κάποια θέματα ε, που μας απασχολούν εδώ στο Κοινοβούλιο θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και πάρα πολύ φιδωλοί όσο και νόμιμοι στη διαχείρισή μας. Βρισκόμαστε στην ετήσια διαδικασία της απαλλαγής και παρά τη ρουτίνο που έχουμε πλέον αποκτήσει σήμερα ε, έχουμε μία πρεμιέρα. Για πρώτη φορά στην Επιτροπή σας καλωσορίζω αξιότιμη κυρία Άστον, είπατε πρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα εξωτερικά ε, ζητήματα. Σας Ευχαριστούμε και χαιρόμαστε που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας. Είναι και ευρύτατο το ερωτηματολόγιο το οποίο απαντήσατε. Ε, είναι στα σκαριά ακόμα η υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Τώρα δημιουργείται με τη συνθήκη της Σαβώνας και αυτό εξηγεί και την πληθώρα των ερωτήσεων που έχει η Επιτροπή μας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας έχουμε ενώπιόν μας και ελπίζουμε και στη διάρκεια της συζήτησης να απαντήσετε αν όχι σε όλες τις περισσότερες ερωτήσεις. Και τώρα στα αγγλικά σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας δίνω αμέσως το λόγο. Μήπως θέλετε καφέ ή τσάι πριν αρχίσετε. Ο εισηγητή θέλει να κάνει κάποια εισαγωγικά σχόλια. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η απαλλαγή της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης εντάσσεται στην έκθεση για τα λοιπά όργανα, οπότε δεν θα πρέπει να έχω εγώ το λόγο, αλλά ο κύριος Τσανέσκι. Μάλιστα. Δεν τον είχα δει δυστυχώ τον κύριο Τσανέσκι. Ζητώ συγγνώμη για την παράβλεψη αυτή. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα πρώτα απ' όλα να καλωσορίσω τους προσκεκλημένους μας σήμερα, την είπατε εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για την πολιτική ασφαλεία και την εξωτερική πολιτική, την κυρία Καλπίν και τον κύριο Μουγκουρούζα. Είναι η πρώτη φορά που ασχολούμαστε με την απαλλαγή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Βαρόνη Άστον για τον τρόπο με τον οποίο απάντησε αυτή και η ομάδα της ε, στο ερωτηματολόγιο και για την θετική και επικοδομητική προσέγγιση που υιοθέτησαν μέχρι στιγμής. Εκτιμάμε ιδιαίτερα το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ε, αναλαμβάνει το καθήκον της με σοβαρότητα. Φυσικά απομένουν κάποια ερωτήματα για τα οποία θα επιθυμούσαμε περισσότερες πληροφορίες. Πρώτα απ' όλα όσον αφορά το οργανόγραμμα της ε, Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης δεν είναι απολύτως ακόμη σαφές ο ρόλος και οι ευθύνε του κ. Βήμωτ, του Γενικού Γραμματέα. Το αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα, ίσως θα μπορούσατε να μας το δώσετε περισσότερες λεπτομέρειες γι' αυτό. Επίσης το ερωτηματολόγιο είχα ζητήσει συγκεκριμένα, είχα ρωτήσει για συγκεκριμένα μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν καλύτερες συνέργειες μεταξύ της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και της ΔΕΦΚΟ και μεταξύ της EEAS και των Εθνικών Διπλωματικών Αντιπροσωπιών. Έχετε δώσει αρκετέ πληροφορίες, αλλά θα ήθελα να μου επισημάνετε ένα ή δύο πρακτικά μέτρα που έχουν ληφθεί ώστε να διασφαλιστούν οι συνέργειες μεταξύ αυτών των υπηρεσιών. Όσον αφορά την ερώτησή μου που αφορούσε την αυτοαξιολόγηση συμμόρφωσης του IC, ήθελα να μάθω κατά πόσο επανορθώθηκε η κατάσταση και κατά πόσο θα ήταν δυνατόν οι υπηρεσίες σας να μας παρέχουν αυτή τη στιγμή τις δηλώσεις αυτές που έλειπαν. Επιπλέον μπορώ να κατανοήσω απόλυτα τις δυσκολίες διαχείρισης των προμηθειών και των αντιπροσωπιών, της φορολόγησης των αντιπροσωπιών, ειδικότερα σε περιοχές ε, όπου η κατάσταση είναι εντελώς διαφορετική από ε, αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα μπορούσατε να μας παρέχετε κάποιες πληροφορίες όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕΔ προσπάθησε να αλλάξει τις βελτιστές πρακτικές και να μάθει περισσότερα από τις εθνικές πρεσβείες ε, στη μέρη αυτά. Αναφέρατε ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ε, οριστικοποιεί τώρα ένα μνημονίο συνεννόησης με την Όλαφ ώστε να υπάρξει σταθερή συνεργασία. Ε, συνεργασία σε σταθερή βάση. Τι εννοείται με τη σταθερή βάση, τι θα καλύπτει αυτό το μνημόνιο. Υπάρχει κάποια διαδικασία χειρισμού των παραπώνων ε, σε επίπεδο EUMS, INSEN και στην ε, ε, αίθουσα στην αίθουσα πώς αυτά θα λειτουργούν αναφέρατε ότι Πώς θεωρείτε ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτή η διαδικασία χειρισμού των παραπώνων όσον αφορά την ερώτηση για τους ειδικού ε, ε, αντιπρόσωπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είπατε ότι η ΕΣΑΡ είναι υπεύθυνη για την ε, υλοποίηση της εντολής. Μπορείτε να μας πείτε πόσο λεπτομερείς είναι αυτές οι εντολές. Θα μπορούσατε να αναλύσετε λίγο περισσότερο το περιεχόμενο αυτών των εντολών. Όταν σας ρωτήσαμε για τους κατόχους θέσεων από θεσμικά όργανα και τα κράτη-μέλη, κάνατε διαχωρισμό μεταξύ μονίμων και ε, προσωρινών υπαλλήλων. Αυτό σημαίνει ότι οι μόνιμοι προέρχονται από τα θεσμικά όργανα και οι προσωρινής απασχόλησης από τα κράτη-μέλη ή από άλλους οργανισμούς. Όσον αφορά το συνολικό ποσοστό εκτέλεσης ε, του προϋπολογισμού 2011, μας ενημερώνεται ότι δεν ήταν ε, δυνατό να το παρέχετε για το 2011 λόγω κάποιων δεσμεύσεων. Ωστόσο, θα έπρεπε τουλάχιστον να μπορούσατε να μας δώσετε έναν υπολογισμό κατά προσέγγιση. Είναι δυνατόν να μας το παρέχετε. Τέλος, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εκ των προτέρων, κυρία Άστον, για τις απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Τσανέσκη ως ε, εισηγητής ε, της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού ε, του Κοινοβουλίου για αυτό το τμήμα του προπολογισμού. μιλήσατε και τώρα καλό είναι να έχει σύντομα τη δυνατότητα να τοποθετηθεί και το ελεγκτικό συνέδριο δεδομένου ότι η κυρία Άστον κατά τις 10 θα πρέπει να αποχωρήσει λόγω άλλων ανηλμένων υποχρεώσεων έχει μια πτήση να προλάβει ε, θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε με τον Chief Executive Officer ε, Sullivan. Ο κύριος Κάρελ Πίνξτεν έχει το λόγο παρακαλώ από το ελεγκτικό συνέδριο πριν την κυρία Άστον. Ε, ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πάρα πολύ χαιρόμαστε που είσαστε εδώ και κάνουμε αυτή την πρεμιέρα. Και έχουμε εδώ την παρουσία τριών συναδέλφων από το ίδιο συνέδριο. Ο συνάδελφος κύριος Τομέ Μουγκουρούθα εδώ παρίσταται γιατί εκείνος ήταν ο βασικός συζητητής για το διοικητικό τμήμα της απαλλαγής. Επίσης εδώ παρίσταται ο κύριος Φαζάκας γιατί εκείνο πρόκειται να είναι ο βασικό συγκριτή για τον οικονομικό έλεγχο που θα γίνει τώρα επί τη ΕΕΔ. Οπότε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μα προσκαλέσατε και θα ήθελα να ξεκινήσω με κάποιε προσαγωγικέ παρατηρήσει και στη συνέχεια να ασχοληθούμε με την ετησία έκθεση για τη χρήση του 11 και κατά τρίτο θα ήθελα να διατυπώσω κάποιες καταληκτικές παρατηρήσεις και ξεκινάμε λοιπόν με τα εισαγωγικά σχόλια. Πρώτα πρώτα θα πρέπει να σας πω ότι με μεγάλη μου ικανοποίηση είδα στην σελίδα 28, συγγνώμη, 38 της ε, έκθεσης δραστηριοτήτων του, της χρήσης του 11 της ε, ότι εκεί θέλετε τέλος πάντων προτίθεστε ε, να βρίσκεστε σε πλήρη λειτουργία της υπηρεσίας σας περί τα μέσα του 2013. Αυτά είναι καλά μαντάτα και για μας γιατί ε, ακριβώς αυτό συμβλέει με το, το, το, πρόγραμμα του ελέγχου μας. Οπότε, έχουμε αυτά τα πρώτα έτη δραστηριότητα που αυτό ήταν κάτι σαν βάπτισμα πυρός για την ΑΕΔ. Είχαμε την Αραβική Άνοιξη, τις συνέπειές τους κλπ. κλπ. Οπότε θεωρώ ότι η εκπρόσωπος ε, προσδοκά να υπάρχουν λιγότερο έντονες Εκδηλώσει στη συνέχεια τη δραστηριότητα, τέλο πάντων έχουμε και άλλα που πρέπει να γίνουν. Θα πρέπει να γίνουν προσλήψεις και θα πρέπει επίσης να υπάρξει μια αποτελεσματική ε, σχέση με την αντίστοιχε αντίστοιχες και γενικές διευθύνσει, Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ βασικό για μας ε, ως ε, ελεγκτέ. Ήδη, όπω σα έχω πει, κυρία Άστον, λέει διάστον ότι είναι πάρα πολύ βασικό αυτού του είδους οι αρμοδιότητες, εκείνες δηλαδή που είναι κοινέ ε, για την ΕΕΔ και την ΤΕΒΚΟ, θα πρέπει να είναι πάρα πολύ σαφές. Και γι' αυτό και το Ελεκτικό Συνέδριο είναι πεπισμένο ότι θα πρέπει η αναπτυξιακή βοήθεια να είναι υψηλή ποιότητα και αυτό θα πρέπει να καλύπτει όλου ε, όσου εμπλέκονται σε αυτό. Τώρα, ε, ακούσαμε και λάβαμε υπόψη για αυτά τα οποία είπε ο εισηγητή κ. Τσαρνέσκη. Τώρα για να δούμε τι γίνεται με κάθε αυτή την αναπτυξιακή έκθεση του 2011. Για να το δούμε σε δυο αξονε άξονες. Πρώτα-πρώτα όσον αφορά τι διοικητικέ δαπάνε. αυτό που εμείς ε, το έχουμε εντάξει στο ένατο κεφάλαιο της δικής μας εκθέσεως και επίσης κάποιες άλλες ε, παρατηρήσεις για την για στις παραγράφους 9 εδάφη 25 και 9 εδάφη 28 και έχουμε επίσης έχουμε και το κεφάλαιο 7 ε, για την ε, διεύρυνση οπότε όσον αφορά πάλι αυτό τον πρώτο άξονα όσον αφορά τις διοικητικές δαπάνες της ΕΕ και το κεφάλαιο 9 λοιπόν στις δικές μας έκθεσεις εδώ πάλι ε, χωρίζεται αυτό το τμήμα σε άλλα δύο. Πρώτα-πρώτα του ανθρώπινου πόρου και στη συνέχεια τους ε, διαγωνισμούς. Όσον αφορά επομένω την ε, διαχείριση του προσωπικού, έχουμε εδώ δύο προβλήματα που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Όπω βλέπετε στο κείμενο, στο κεφάλαιο του 9, σε 6 από τι 17 περιπτώσεις ελέγχων δεν είχαμε επικαιροποιημένα στοιχεία που αφορούσαν την οικογενειακή προσωπική κατάσταση των μελών του προσωπικού. Οπότε και ε, κατά συνέπεια δεν εκταμιεύθηκαν οι πόροι που θα έπρεπε για αυτά τα πρόσωπα. Επίσης, είχαμε κάποιες ε, συμβάσεις προσλήψεως προσωρινού χαρακτήρα που υπογράφηκαν τρεις με επτά μήνες αφού άρχισαν να δουλεύουν αυτά τα πρόσωπα. Και μιλούμε για τρεις από τις οκτώ περιπτώσεις που ε, έχουμε εξετάσει. Επίσης, ε, έχουμε μια συγκεκριμένη περίπτωση. Έχουμε ένα, μια σύμβαση για υπηρεσίες ασφαλείας στη Βενεζουέλα που υπάρχει 24 χρόνια και δεν έχει τροποποιηθεί, κάτι το οποίο το διαφωνίζουμε στην παράγραφο 9 και 27. Στη συνέχεια δε, έχουμε ε, κάποιες ε, ελλείψεις οι οποίες παρατηρούνται σε όλη την ε, διαδικασία των συμβάσεων και διαγωνισμών όσον αφορά την σύναψη τέτοιων συμβάσεων υπηρεσιών ασφαλείας. Επομένως, τα προβλήματα είναι σε σχέση με τους ανθρώπινους πόρους, το προσωπικό δηλαδή και τους διαγωνισμούς και συμβάσεις προμήθειας. Επίσης, έχουμε τώρα Έχουμε τώρα το κεφάλαιο 7 και επίσης είναι της που αφορά δραστηριότητε για τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Ανάπτυξη, παριθμών 8, 9 και 10. Φαντάζομαι θα θυμάστε ότι κατά την πρόσφατη ακρόαση του Επιτρόπου Πίμπαλς ε, είχαμε σταθεί στη συζήτηση που έγινε για την ε, έκθεση του 2011 στο κεφάλαιο 7, στο κεφάλαιο επίσης για το Ταμείο Ανάπτυξης διότι υπήρχαν και κάποιες παρατηρήσεις που, έχουν, που ισχύουν και για την ΑΕΔ. Και η προγραμματιστή βοήθεια για τις χώρες εταίρους μας είναι κάτι που αποτελεί κοινή ευθύνη, κοινή αρμοδιότητα ΤΕΒΚΟ και ΑΕΔ. Οπότε, τα σχετικά ποσά και οι μηχανισμοί παροχής της αναπτυξιακής ε, βοήθειας έχουν καθοριστεί. Και αυτό φυσικά καλύπτεται, αυτό το ποσά καλύπτεται τον προπολογισμό. Οπότε να δούμε τώρα, υπάρχουν κάποια προβλήματα σχέση με την ε, υποστήριξη, την κάλυψη από τον προπολογισμό. Έχουμε τώρα στο κεφάλαιο 7 δύο παραγράφους, 9 και 10. Και όσον αφορά τις δύο παραγράφους επίσης, τις έκθεσεις για το Ταμείο. Πρώτα-πρώτα, αυτή η κάλυψη του προπολογισμού ε, σχετίζεται με κάποια αδύναμα, με κάποια ελλειπή συστήματα διαχείρισης των δημοσίων πόρων. Επίσης, η, ο οικονομικός σταματά σε ένα, συγκεκριμένο, σε ένα συγκεκριμένο στάδιο, όταν δηλαδή έχει γίνει η μεταφορά των πόρων. Επίσης, ε, εδώ πέρα έχουμε μια ευρύ ερμηνεία, για να το πω διπλωματικά, σχέση με το ποιος είναι ο επιλέξιμος. Οπότε, θα πρέπει στα σοβαρά να δούμε κατά πόσον αυτοί οι κίνδυνοι που υπάρχουν είναι κάτι που θα πρέπει να θεωρηθεί απαράδεκτο ή όχι σε σχέση με τον Ευρωπαίο φορολογούμενο. Διότι όλη αυτή η κατάσταση και κυρίως οι, οι ελληπείς διαδικασίες και συστήματα διαχείρισης των δημοσίων οικονομικών είναι κάτι το οποίο ε, επιδέχεται ή οδηγεί σε διαφθορά και απάτη. Και όπως είπαμε και θα σας και ο κ. Φαζάκας θα, συζητήσει τα θέματα αυτά τα οποία επίσης όσον αφορά την, την πλήρη λειτουργία της ΕΕΔ είπαμε ότι θα γίνει μέχρι τα, τα, τα μέσα του τρέχοντος έτους. Οπότε, εν κατακλείδη, θα ήθελα να σας πω ότι αν έχετε κάποιες ερωτήσεις για το κεφάλαιο 9, μην διστάσετε. Ο Ισπανός συνάδελφος κύριος το Μουγκούρθα θα σας ε, καλύψει, ελπίζω, κάθε σας ερώτηση. Ευχαριστώ κύριε Πίνξτεν ε, για την τοποθέτηση του ελεκτικού συνεδρίου και τώρα θα πρότεινα να δώσουμε το λόγο στην κυρία Άστον για να μας ε, κάνει την παρουσίασή της για να απαντήσει στη συνέχεια στις ερωτήσεις μας. Συγκεκριμένα των εκπροσώπων των πολιτικών ομάδων. Έχετε το λόγο. Κάνω την αναρκτήρια παρατήρηση και θα απαντήσω σε νέα ερωτήσεις του κύριου Τζανέσκη και κατόπιν θα απαντήσω και στα όσα είπε ο κύριος Πίνστεν από το Ελεκτικό Συνέδριο. Μεγάλη μου χαρά με εδώ στην συνεδρία σα και σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εσά και την Επιτροπή σα, διότι ε, οργανώσατε αυτή την ε, συνάντηση ε, και καταφέραμε να, βρούμε τον χρόνο μια που και εγώ έχω τόσε πολλέ υποχρεώσει και ελπίζω ότι καλύψαμε, θα μπορέσουμε να καλύψουμε τώρα πάντων 137 ερωτήσει και θα γίνει τελικά ο κατάλληλο διάλογο και εδώ και μετά από αυτή τη συνεδρίαση. Οπότε μεγάλη μου χαρά παρίσταμε στη συνεδρίαση όπως προείπα, διότι περιμένω πώς και πώς τις δικές σας ιδέες και προτάσεις, γιατί αυτό που προσπαθώ να κάνω είναι να δούμε πώς θα μπορέσουμε να έχουμε την οικονομική διαχείριση τη, τη διοίκηση, να κάνουμε ό,τι, ό,τι χρειάζεται, τόσο να μπορέσουμε ως ΕΙΕΔ να κάνουμε τη δουλειά μας, γιατί αυτό που χρειάζεται είναι να υπάρχει η αναγκαία ευελιξία, γιατί ε, οι προκλήσεις είναι πάρα πολύ σημαντικές. Έχουμε ε, όχι μόνο τις εντυπωσιακέ αλλαγές εδώ στη γειτονιά μας, αλλά έχουμε και επίσης την οικονομική δύσκολη συγκυρία. Και επίσης έχουμε ε, Επομένως αυτό το δύσκολο πλαίσιο, γιατί αυτό το οποίο πρέπει να γίνει είναι να συνεργαστούμε για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε όσο γίνεται καλύτερα τους περιμένους πόρους που έχουμε και να μπορέσουμε να πετύχουμε τους σκοπούς που έχει τάξει για μας η συνθήκη της Λισαβόνας. Βεβαίω και θεωρώ είναι πάρα πολύ θετική συνεχής υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, για την πολιτική μας, για όλους τους τομείς πολιτικής μας και όπως ε, είπατε κύριε Πρόεδρε θα πρέπει κάτι να κάνουμε για αυτές τις ε, αλλαγές που έχουν γίνει για την ε, Αραβική Άνοιξη. Θα πρέπει να δούμε πώς θα αναβαθμίσουν την πολιτική γειτονία, να έχουμε μια task force, μια καινούργια αντίληψη για αυτήν, ούτως ώστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο άμεσα να εμπλέκεται και έτσι να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις αλλαγές σε κάθε τομέα. Επίσης θα πρέπει όλο ένα και περισσότερο να αντιμετωπίσουμε τις ε, κρίσεις όταν ε, επίσης και να μην ξεχνούμε τι γίνεται στο κέρα της Αφρική της Σομαλία, αλλά και στο Σαχέλ, όπως επίσης και τις δρομικές εξελίξει στη Συρία. συνεχίζουμε τα μεταβολές σε όλο τον ε, κόσμο, Μπούρμα, Μιανμάρ, οπότε έχουμε τώρα όλες αυτές τις εξελίξεις και δεσμές μας για την Μέση Ανατολή. Επομένως, ε, ε, έχουμε πρωταγωνιστικό ρόλο στις συνομιλίες με το Ιράν, στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Πριστίνα και Βελιγραδίου, οπότε ε, έχουμε τους βασικούς μας στρατηγικού εταίρου, με του οποίου έχουμε δεσμευτεί μαζί να αντιμετωπίσουμε αυτέ τι προκλήσει. σε μια καινούργια, ένα καινούριο πλαίσιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, κάτι το οποίο διαπνέει κάθε σχέση ε, που έχουμε με οποιαδήποτε χώρα παντού στον κόσμο, οπότε πολλά έχουν πολλά παραδείγματα που να σας πω, οι περισσότερα, μεγάλη λίστα από, από, από στόχους, έχουμε την προστιθέμενη αξία που δίνουν οι πολιτικέ και τα θεσμικά τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να μπορούμε να έχουμε μια συμβολή με καλή σχέση κόσμου. Αποτελέσματο για τι εξωτερικέ μα σχέσει και όλα αυτά έχουν να κάνουν βέβαια με το πόσο μπορούμε να έχουμε μια προσέγγιση τέτοια η οποία να μπορεί να καλύψει ε, αυτή μας την πολιτική με τα κατάλληλα μέσα πολιτικής, εργαλεία, ό,τι υπάρχει και ό,τι μπορεί να γίνει και σε εθνικό επίπεδο. Αλλά αυτό χωρίς να έχουμε επικαλύψεις. Οπότε να έχουμε αυτήν την προστιθέμενη αξία. Οπότε μέσα σε αυτήν την οικονομική συγκυρία αυτό το οποίο επιζητούν ολοένα και περισσότερα κράτη-μέλη είναι την βοήθεια από την ΑΕΔ και βέβαια έχουμε σε αυτές τις 140 περίπου αντιπροσωπείες παντού σε όλο τον κόσμο οπότε και εμείς βέβαια ε, διαπόμαστε από το ίδιο οικονομικό πλαίσιο, περιορισμούς, γι' αυτό και θα πρέπει να αξιοποιήσουμε όσο γίνεται καλύτερα ε, τους πόρους που διατίθενται για μας. Ό,τι προβλέπεται από το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έγιναν ε, δύο έλεγχοι, να δούμε πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα πάνε, να μην έχουμε επικαλύψεις με, με τα θεσμικά όργανα και 10% των θέσεων αφορούν τη, τη καινούργια διοργάνωση, τη οργάνωση μάλλον, ε, να δούμε τι θα κάνουμε για τους τομείς εθνικής άμυνας και εξωτερικών και να δούμε πώς θα καλύψουμε τις ομάδες του Συμβουλίου ούτως ώστε τελικά να μπορούμε να λειτουργήσουμε αυτόνομα. Επίσης, έγινε ακόμα ένας, ένας ε, έλεγχος ούτως ώστε να δούμε πώς θα μετακινήσουμε κάποιους από τους υπαλλήλους μας από, το, από την έδρα μας εδώ στις αντιπροσωπείες. Γιατί άλλο οι δικέ μα αντιπροσωπείε και άλλο οι παλαιότερε που είχε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οπότε γι' αυτό σε τέτοιου ταραγμένου καιρού θα πρέπει να μπορεί το προσωπικό μας να, αναδρά άμεσα από άμεσα έχουμε κάποια κρίση. Βέβαια υπάρχουν και πολλοί κίνδυνοι ε, και ας πούμε ε, τι συνέπειες έχουν οι πράξεις μας, αλλά επίσης πώς και θα λειτουργεί με ασφάλεια η κάθε μας αντιπροσωπεία. Γιατί μιλούμε τώρα για κάποιες πάρα πολύ δύσκολες στιγμές, ε, επικίνδυνα μέρη, δεν λειτουργούν τα πράγματα το ίδιο παντού, οπότε θα πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε να δανειστούμε τις άριστες πρακτικές από την εμπειρία ε, από, τις άλλα, τα άλλα θεσμικά όργανα και όσον αφορά τους οικονομικούς ελέγχους αυτό ε, ισχύει και γι' αυτό και είναι θετικό το ότι ήρθε εδώ το ελληνικό συνέδριο και πώς θα, τελικά θα ολοκληρώσουμε και το μνημόνιο κατανόησης σε συνεργασία με την Όλαφ. Έχουμε καινούριε διαδικασίες πάντως, καινούργια χαρακτηριστικά που διέπουν το έργο μας επίσης και το πώς θα έχουμε παράλληλα κυκλώματα ελέγχου των οικονομικών, ε, επίσης καινούργια πολιτική προσλήψεων ε, των αποσπασμένων διπλωματών από τα κράτη-μέλη. Άλλος στόχος αυτός, οπότε και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Θα πρέπει να συνεργαστούν τα κράτη-μέλη, θα πρέπει να δούμε πώς θα επηρεάσουμε το καινούργιο πνεύμα συνεργασία, τη καινούργια κουλτούρα συνεργασία. Αλλά πάντω η ΕΔ επίση ε, συνεργάζεται πάρα πολύ στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα άλλα θα συγκαρούν. Επίσης έχουμε και την δήλωσή μας για την απόδοση ευθυνών. Επίσης ε, ε θα πρέπει να δούμε πώς θα έχει συνέβη η εξωτερική μας πολιτική ε, και όσον αφορά την, την οικονομική βοήθεια, ε, συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις λειτουργικές δαπάνες και για το πώς θα γίνει η διαχείριση όλων των ε, που αφορά τις αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πάντως Ντέβιτο ε, Σάλβαν που είναι ο βασικός μας ε, εκτελεστικός διευθυντής έκανε μια έκθεση και εκεί πέρα είδαμε ότι ε, έτσι θα μπορούσαμε να διαχειριστούμε τον προπολογισμό. Και έτσι θα συζητήσουμε και θα δούμε τι γίνεται με τον προηγούμενο του 2011. Οπότε θα βρούμε τον τρόπο για να μπορεί να έχει εμπιστοσύνη σε εμά, ο βέβαιο φορολογούμενος, να πιάσουν τόπο τα χρήματα τα οποία πληρώνει κατά κάποιο τρόπο, μια που είναι πάρα πολύ συγκεκριμένε οι ευθύνε μας, οι αρμοδιότητέ μας, αλλά μην μη γελιάστε, εμείς ε, θέλουμε να είμαστε υπεύθυνοι, να είμαστε υπόλογοι, να κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο. Για να δούμε τώρα μερικά από αυτά τα οποία είπε ο κύριος ε, Τσερνέσκι. Να απαντήσουμε εντάξει ότι του πρώτο πρώτο μας είπατε τι γίνεται όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, το, το αρχικό. Και αυτός ο γενικός διοικητικός διευθυντής συντονίζει. Επίσης, ασχολούμαι κάποια πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Σήμερα, ας πούμε, ασχολείται με τα όσο γίνονται στην Σύρια. Προεδρείε. Πρόκειται με τον πρώτο συμβουλίο να πάει επίσης στην ε, Αίγυπτο, σε αμέσως πόνες εβδομάδες. Επίσης, προσπαθεί να εξασφαλίσει κάποιο είδους στρατηγική συνέπεια στη δράση μας. Αυτά για τον David Σάλιβαν ε, που συνεργάζονται. Οπότε καλύπτεται όλος ο φορέας από τα διοικητικά, διαχείριση προσωπικού μέχρι τις στρατηγικές, τα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Πολύ, κάτι πολύ σημαντικό τόσο ώστε να προωθηθεί ο ρόλος της υπηρεσίας μας αλλά και του Συμβουλίου αλλά βέβαια και με τον ε, ρόλο μας Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Επίσης, είπατε για την Ντεύκο, για τη συνεργασία μας. Ένα καλό παράδειγμα είναι το τι γίνεται στο κέρας Αφρικής. Με το που συγκροτήθηκε αυτή η υπηρεσία, για πρώτη φορά προσπαθήσαμε να οργανώσουμε, να, επιστρατεύσουμε το προσωπικό από παντού από όλα τα θεσμικά όργανα, η αναπτυξιακή βοήθεια, ανθρώπινα δικαιώματα κλπ. Και όλα αυτά ήταν πάρα πολύ χρήσιμα για το μέλλον της ε, Σομαλίας. Και σε συνεργασία με όλες τις ε, χώρες της περιοχής είπαμε να εξασφαλίσουμε την ε, θαλάσσια ασφάλεια, να βρούμε εναλλακτικέ για τους νέους, ούτως ώστε να μην γίνονται πειρατές, να βρούνε κάποια δουλειά. Και όλα αυτά, όλα αυτά αφορούν το μέλλον της χώρας. Επομένως, η ΕΕ δεν μπορεί παρά να συνεργάζεται με την ΔΕΒΚΟ. Εδώ, στις Βρυξέλλες. Και θα μπορούσα να σας πω άλλα 20-30 παραδείγματα τέτοια. Πρόκειται για μια συνέργεια. Αυτό γίνεται. Βέβαια, δυνάμει τη εντολή που έχουμε, αλλά όλα αυτά με ένα σφαιρικό τρόπο για να καλύψουμε με αποτελεσματικό τρόπο τα καθήκοντά μας. Αυτό αφορά και την διεθνή διπλωματία για τις χώρες που βρίσκονται εκεί στο κέρας Αφρικής, είχα πάει τον Αύγουστο στο Μογκαντήσου, οπότε και όλες οι εμπλεκόμενες χώρες μέλη ήταν συνομιλητές μου. Θέλαμε να δούμε αν έχουμε ό,τι χρειάζεται, ούτω ώστε να αντιμετωπίσουμε την πειρατεία. Κοινέ ναι, ήταν οι αρχές που διέπνουν αυτές τις προσπάθειες. Συντονισμός και συνέργεια. Να, Πήγαινε και απευθυνθείτε στου πρέσβει των χωρών μελών. Τι έγινε στο κέρας Αφρική και όλοι θα σα πούν ότι αυτό ήταν παράδειγμα προ μίμηση. Δεν είπα πάρα πολύ καλό παράδειγμα συνέργεια, συνεργασία. Είπατε επίση για αυτά τα ποσά τα οποία έλειπαν. Βέβαια μπορούμε να σα τα παράσχουμε. Άρθρες πρακτικέ, εμπειρία από τις ε, πρεσβείε κρατών μελών. Προσπάθησα αυτό να σου το πω στην εισήγησή μου. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, να, να επιστρατεύσουμε αυτούς τους διπλωμάτες με την εμπειρία τους. Η ομάδα η οποία διαχειρίζεται τα όσα κάνει κάθε μας αντιπροσωπεία, όλα αυτά τα δύσκολα που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό και έχουμε ε, κόσμο και προσωπικό και διπλωμάτες και από την Κομισιόν από παντού, από παντού. Και είναι πολύ ενδιαφέρον το να έχει κανείς α, αυτή την πανσπερμία προσωπικού και ταυτόχρονα να προσπαθούμε να ακολουθήσουμε αυτές τις άριστες πρακτικές για τις οποίες φημίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανταλλαγή πληροφοριών, ε, πρόσβαση σε έγγραφα, να καθορίσουμε, να οριοθετήσουμε τη σχέση με την Όλαφ, θεσμική μας σχέση, οπότε από τα αποτελέσματα θα κρίνεται. Και αυτό το situation room, αυτή την ε, αίθουσα επιχειρήσεων, ούτως πίνω. Ε, πρόκειται για ε, αίθουσα επιχειρήσεων, ας πούμε, που λειτουργεί κάθε μέρα όλο το χρόνο. Μέρα και νύχτα. Θέματα τα οποία αντιμετωπίζονται. Κρίσεις, κατεπήγοντα, συνεχή συμπληροφορία. Οπότε και γι' αυτό και α πούμε παρακολουθούμε τι γίνεται στην Πριστίνα, στο Βελιγράδι. Πολύ στενή είναι η συνεργασία. Οπότε και αυτόν τον τρόπο ε, κάνουμε κάτι το οποίο δεν ίσχυε προηγουμένως και επομένως αυτό είναι πολύ βασικό και η γλώσσα όπω είπατε έχει τέτοιο προσωρινό χαρακτήρα συνεργασία με του διπλωμάτε, οπότε ο ό,τι λείπει έχετε δίκιο θα σας δώσουμε ό,τι στοιχεία χρειάζονται το, το είπαμε αυτό έτσι έτσι πρέπει να γίνει Α, να βάλω εδώ τελεία αυτά για τον κύριο Τσαρνέτσκι τώρα κάτι για το κείμενο και για τα όσα είπε μάλλον πάντων ο κύριος Πίνγκστον Ήταν πολύ σημαντική η επίσκεψή μου στο ελεγκτικό συνέδριο. Πιστεύω ότι το, ο αρμόδιος ε, ασχολήθηκε με αυτό το πρόβλημα και το διόρθωσε. Όσον αφορά το έκτακτο προσωπικό, το εξηγήσαμε. Στην αρχή τη υπηρεσία χρειάστηκε περισσότερος χρόνος. Εγώ θυμάμαι ότι υπέγραφα πράγματα κάποιες μέρες και ήμουν η μόνη που μπορούσα να κάνω τη δουλειά. Δεν υπήρχε αρκετό κόσμο και τώρα έχουμε εγκαθιδριστεί σωστέ διαδικασίες και ζητώ συγγνώμη για όσους δεν έλαβαν τη συμβάση του όσο γρήγορα έπρεπε. Έχει διορθωθεί τώρα η κατάσταση. Τώρα, όσον αφορά τη δημοσιονομική στήριξη, είχαμε μια συναρπαστική συζήτηση γι' αυτό στο Λουξεμβούργο όταν είχα έρθει. Ε, έχουν γίνει διάφορα συζητήσει επί του θέματο. Πολλέ χώρε λένε χρειαζόμαστε βοήθεια για να οικοδομήσουμε ικανότητες εντός της κυβέρνησης ώστε να μπορεί να λειτουργεί από μόνη της ο τομής υγείας, εκπαίδευσης, παιδείας, δικαιοσύνης, οτιδήποτε. Και μετά λέμε ότι όταν λειτουργούμε εκτός κυβέρνηση και δίνουμε χρήματα κατευθείαν σε μη κυβερνητικούς οργανισμού ή σε άλλες υπηρεσίες, δεν βελτιώνουμε το έργο αυτό εμείς. Δηλαδή πρέπει να κάνουμε κάποια εξισορρόπηση διότι εξορισμού πολλές χώρες που χρειάζονται δημοσιονομική στήριξη δεν έχουν τις ικανότητες που θα επιθυμούσαμε να έχουν. Ήταν πολύ σωστή η παρατηρήσή σας. Πρέπει να είμαστε απολύτως σαφείς στις διαδικασίες αυτές. Γι' αυτό το λόγο το Σεπτέμβριο του 2012 εκδώσαμε κατευθυντήρες γραμμές που θα εξετάζουν, θα αντιμετωπίζουν καλύτερα τη διαφάνεια και παροτρύνουμε και τα κράτη-μέλη να κάνουν το ίδιο ώστε να διασφαλίσουμε ότι θα μπορέσουμε να οικοδομήσουμε σωστά αυτέ τι ικανότητε. Έχουμε μεγάλε προκλήσει σε χώρε όπω το Πακιστάν, το Αφγανιστάν. Έχουμε μιλήσει εκτενώ με αυτού ε, όσον αφορά το πόσο επιθυμούν να ε, υλοποιηθεί κάτι τέτοιο και πόσο μπορούν. Αλλά φυσικά η προστασία των κονδυλιών είναι σημαντική. Είναι ένα ζήτημα στο οποίο πιστεύω ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε τη δημοσιονομική στήριξη και να βοηθήσουμε αυτές τις χώρες να αναπτύξουν τα απαραίτητα μέσα ε, στο πλαίσιο της ασφάλειας φυσικά ε, και της διασφάλισης ότι ξέρουμε πού πηγαίνουν τα χρήματα αυτά. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Άστον που απαντήσατε αυτές τις ερωτήσεις και τώρα δίνω το λόγο για τον πρώτο κύριο συζητήσεων και περιορίζω το χρόνο ομιλίας του καθεμιλητή σε δύο λεπτά. Κάθε ομάδα λοιπόν θα έχει την ευκαιρία να κάνει μια ερώτηση. Πρώτα απ' όλα η Γκέγκρέσκε από το ΕΛΚΑ, δεύτερη σοσιαλιστές. Ποιος θα μιλήσει για τους σοσιαλιστές. Ο κ. Κάλφιν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, θα ήθελα να πω ότι με την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης είχαμε πρωτοφανή διαφάνεια. Αλλά αυτό δεν πιστώνεται στην ίδια την υπηρεσία εξωτερικής δράσης, από το σχεδιασμό της ήταν έτσι. Για τα έγγραφα του προπολογισμού, ο τρόπος με τον οποίο στήθηκε η ίδια η υπηρεσία, το φροντίσαμε από την αρχή και το αναγνωρίζω αυτό. Έχουμε πλέον ε, μια τεχνογνωσία για τη ε, διαχείριση και ε, των οικονομικών ζητημάτων και τα λογιστικά και το θέμα των έξυπνων οικονομιών, το smart savings. Δεν είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη όμως με τις απαντήσεις που δώσατε στο ερωτηματολόγιο. Οι διαγωνισμοί ε, που προκυρήσετε, τι κοστίζουν. Ε, είναι 8.800 υποψήφοι, 1.300 οι συνεντεύξεις. Ε, το εκτιμώ πάρα πολύ. Είναι βαριές οι διαδικασίες, είναι αξιόλογοι οι άνθρωποι, αλλά όταν η θέση είναι 181 είναι πάρα πολύ κακό αυτό για 181 θέσεις. Και τα κράτη-μέλη επιλέγουν 40% των πρέσβεων και των, στις αντιπροσωπείες ε, είναι από ε, τα Υπουργεία Εξωτερικών. Μα είχαμε συνεννοηθεί για ένα τρίτο. Γιατί έγινε αυτό 40%. Ε, στη συνέχεια, τι κάνετε για τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης. Είναι μεγάλη απουσία του δικού μας προσωπικού ε, των ευρωπαϊκών κοινοτήτων στις τρίτες χώρες. Αντιπροσωπείες, τι κάνετε γι' αυτό, είναι ακόμα ανοιχτή υπόθεση ή θεωρείτε ότι πρέπει να γίνει ε, κάτι γι' αυτό. Ανταλλαγή απόψεων επίσης με τα κράτη-μέλη στις τρίτες χώρες. Στην ερώτηση 131 απαντάτε κανένα πρόβλημα. Μα εγώ μιλάω με τους πρέσβεις και όλοι ανεξαιρέτως μου λένε ότι δεν έχουν δει ούτε ένα χαρτί από τα κράτη-μέλη. Αυτοί καλούνται να τα στέλνουν όλα, αλλά δεν του απαντάνε. Εσεί καλό είναι να μα λέτε ότι δεν υπάρχουν προβλήματα. Μήπω υπάρχουν και δεν το γνωρίζετε και πώ μπορούμε να υποστηρίξουμε. Σαν το Μεξικανικό στρατό έχουμε γενική διεύθυνση με 44 άτομα, διεύθυνση με 22. Τι οργάνωση είναι αυτή ε, στο αρχηγείο σας. Ε, μπορείτε να διαμορφώσετε καλύτερα την κατάσταση για να υπάρχει και συγκρίσιμη κάπως ε, ε, λειτουργία στις διευθυντικές θέσεις με άλλα θεσμικά όργανα. Ευχαριστώ κύριε Γκρέσλε. Κύριος Καλφίν από Σοσιαλιστές και Δημοκράτες για δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω κυρία Αστόν για τις ε, πλήρε απαντήσεις που δώσετε στις ερωτήσεις που κάναμε προς σας. Έχω δύο ερωτήσεις όσον αφορά το συντονισμό με άλλους ε, παράγοντες ε, στις διάφορες χώρες. Αναφέρατε στη Σομαλία όπως και σε άλλες περιπτώσεις έχετε ένα πολύ καλό μηχανισμό συντονισμού των δραστηριοτήτων με άλλες υπηρεσίες ε, όπως την ΔΕΦΚΟ, θα συμπεριλαβώ και την αρρωγή εκτακτής ανάγκης αλλά και με άλλους ε, συμμετέχοντες εθνικούς, διμερείς κτλ. Τι θα γίνει ώστε αυτό να αποτελεί πρότυπο, όχι απλά να αναφέρουμε βέλτιστες πρακτικές όπως στην ΚΕΙΝΕ και στη Σομαλία, διότι πολύ συχνά η συμπληρωματικότητα μπορεί να επιφέρει τεράστια προστιθέμενη αξία στο έργο της ε, ΕΙΕΔ. Η δεύτερη ερώτησή μου αφορά τη σύνδεση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας ε, Εξωτερικής Δράσης και των Εθνικών ε, Διπλωματικών Υπηρεσιών. Αναφέρατε ότι έχετε την ποσόστοση του ενός τρίτου του προσωπικού, του απεσπασμένου προσωπικού Πιστεύετε ότι αυτός ο μηχανισμός απόσπασης, επειδή γνωρίζω ότι σε κάποιους τομείς, ε, σε κάποιες περιοχές ε, δεν θέλουν να αποσπάσουν προσωπικό τα κράτη-μέλη για δημοσιονομικό, λόγω δημοσιονομικών περιορισμών. Πιστεύετε πώς θα γίνει αυτό στο μέλλον σε εθνικό επίπεδο. Και τέλος, προβλέπετε κάποιες ε, επιπλέον ιδέες για να παγιώσετε το έργο των εθνικών διπλωματικών αντιπροσωπείων σε θέματα αντιπροσώπευσης καλύτερης χρήσης των κονδυλίων, των ικανοτήτων που υπάρχουν στα... Ε, ώστε να υπάρξουν συνέργειες και να υπάρξει προσθέμενη αξία στο έργο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριος για το χρόνο που τηρήσατε. Ο κύριος Κυλακάκης από του Φιλελευθέρους παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Άστον για την παρουσία σας και την παρουσίασή σας. Θα είμαι πολύ σύντομος γιατί σε δύο λεπτά πρέπει να καλύψω πολύ μεγάλο πεδίο. Πώς αντιλαμβανόμαστε τη δική σας ε, αποστολή. Έχετε 141 αντιπροσωπείες. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η δουλειά σας θα πρέπει να υποπτεύεται τον κόσμο ολόκληρο. Είναι πραγματικά ε, πολύ μεγάλο έργο και θέλω να σας βοηθήσω. Και εμεί θέλουμε από τις απαντήσεις που δώσατε στις ερωτήσεις μας, τι φαίνεται. Είτε δεν υπάρχουν προβλήματα ή ε, ε, παρατυπίες, άρα έχει αλλάξει κατά πολύ η ανθρώπινη φύση σε ό,τι αφορά την υπηρεσία εξωτερικής δράσης, είτε έχουμε προβλήματα αλλά δεν έχουμε ακόμα τις κατάλληλες διαδικασίες για να τα εντοπίζουμε. Και μάλλον αυτό είναι πιθανότερο, καθώς είναι καινούργια υπηρεσία. Και ο κόσμος είναι αφημένο στη μοίρα του παγκοσμίω και λειτουργεί ε, αποκομμένα. Ε, δύο συγκεκριμένα ζητήματα. Το ένα είναι οι διαδικασίες ε, διαπραγματεύσεων. Οι περισσότερες προμήθειες αγορέ γίνονται με διαπραγματεύσει κάτω από 60.000 ευρώ. Σε πολλές χώρες είναι πολλά λεφτά 60.000 ευρώ. Σε πάρα πολλές χώρες, εκεί που λειτουργούμε και εργαζόμαστε. 60.000 είναι μεγάλο ποσό και μπορεί κανείς να προμηθευτεί πολλά. Ε, μπορείτε να μας πείτε ε, λίγα λόγια. Και δεύτερον, σε ό,τι αφορά τις κατοικίες, είδαμε ε, από τις ερωτήσεις μας ότι είναι πολύ ποικίλε αυτές οι κατοικίες των επικεφαλής. Μπορεί να είναι 270 τετραγωνικά στο Χονγκ Κονγκ και 710 στην Τζαμάικα, Φερρυπίν. Ε, έτσι. Ε, αυτό είναι ένα μικρό ανάκτορο, δεν είναι κατοικία πρέσβη. Και τα συμβόλαια ενοικίασης είναι δεκαετή. Μπορείτε να μας εξηγήσετε και τι γίνεται. Μπορείτε επίσης να ιδρύσετε κάποια νέα υπηρεσία, ένα ειδικό επιθεωρητή που θα σας βοηθάει και θα δίνει περισσότερα κίνητρα στους ανθρώπους να είναι πιο προσεκτικοί στη διαχείριση των κονδύλιων, των φορολογουμένων. Ειδικά σε σχέση, ε, ε, έχουμε τέτοιους επιθεωρητές σε πολλά Υπουργεία Εξωτερικών. Ευχαριστώ. Από τους Πρασίνους δεν βλέπω συνάδελφο. Οπότε πάμε στον κύριο Έπινγκ ε, από τους συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές. Δύο λεπτά πάρκα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Άστον, όταν οριστήκατε πρώτη ως επικεφαλής της ΕΕΔ είχατε πει ότι δεν θα επηρεάζει ιδιαίτερα τον προϋπολογισμό αλλά δύο φορές έχετε ζητήσει αύξηση του προϋπολογισμού πρώτον κατά 5,3% το 2012 και τώρα κατά 4% στο τελευταίο σχέδιο προϋπολογισμού. Η ερώτησή μου είναι λοιπόν για ποιον λόγο μιλήσετε για δημοσιονομική ουδετερότητα. Το άλλο σημείο αφορά ένα παράρτημα του εσωτερικού κανονισμού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιτρέπει στην ΕΕΔ να ξοδεύει εκατομμύρια στέλνοντας το προσωπικό της σε εξωτικές τοποθεσίες για ε, διακοπές ως κίνητρα ή ως ε, ανταμοιβή για δύσκολες ε, αποσπάσεις. υπό την τρέχουσα δημοσιονομική κατάσταση των κρατών μελών ίσως ε, είστε υπερβολικά γενναιόδοροι. Από όσο κατάλαβα επίσης η συγχώνευση της Ευρωπαϊ... των υπηρεσιών ε, Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής και Ευρωπαϊκού Συμβουλίου έχει δημιουργήσει τεράστια γραφειοκρατία με αξιωματούχου που να έρχονται. Δεν είμαι λοιπόν βέβαιος ότι ελέγχεται καλά τη διαχείριση αλλά όπως είχα δει με τον... Επειδή τον κύριο Σάλιβαν, ε, είμαι ανοιχτό να δεχτώ εξηγήσει γι' αυτό. Ε, υποστηρίζω την παρατήρηση του κύριου Πινξέν για τη δημοσιονομική στήριξη. Εγώ επικρίνω δημοσιονομική στήριξη. Το θέμα είναι, αφορά περισσότερο την ποσότητα τη αρρωγή και όχι την ποιότητα. Θα σα υπενθυμίσω ότι στην Τινησία η Τινησία κυβέρνηση του κ. Μπέναλη είχε λάβει 60 εκατομμύρια δημοσιονομική στήριξη πριν εγκαταλείψει. Το ίδιο και ο κύριος Μουμπάρεκ πάνω από 100 εκατομμύρια. Κατά κάποιο τρόπο αυτή η δημοσιονομική στήριξη και η πολιτική γειτονία έχουν καταρρεύσει. Θα, είμαι, θα επικρίνω λοιπόν αυστήρα και θα σα ζητήσω να αναθεωρήσετε, να δείτε τι γίνεται με αυτό το φαινόμενο. Ευχαριστούμε κύριε συναδέλφε που τηρήσατε το χρονικό όριο. Ε, από το EFD, κυρία Αντρέασεν, θα θέλατε το λόγο. Για δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Άστον, όταν η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική δράση δημιουργήθηκε, είχε συζητηθεί ότι η ΕΕΔ μπορεί να αντικαθιστούσε τις πρεσβείες των χωρών. Αυτό δεν διασαφινίστηκε ποτέ, αλλά αυτό που βλέπει σήμερα ο κόσμος είναι ότι πράγματι έχει αυξηθεί ο προπολογισμό Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά περίπου 500 εκατομμύρια και ως αντιστάθμισμα βλέπουν εκφράσεις όπως ισχυρότερη δέσμευση στη Μέση Ανατολή. Αυτό το κόστος είναι πολύ υψηλό για τέτοιου είδους αποτέλεσμα. Δεν θέλω να επικρίνω βέβαια, διότι εδώ είναι η πρώτη χρονιά βέβαια της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, αλλά ταυτόχρονα όπως γνωρίζετε Έχουμε να αντιμετωπίσουμε με συνθήκες σε πολλά κράτη-μέλη και ο κόσμος ε, θα το δει αυτό πολύ, θα το εξετάσει πολύ προσεκτικά. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι η ΕΕΔ θα αντικαταστήσει όντως τις πρεσβείες των κρατών μελών ή όχι. Εγώ προσωπικά δεν είμαι υπέρ μια τέτοια ιδέα, αλλά θα ήθελα να ακούσω και τη δική σα απάντηση. Η δεύτερη μου ερώτηση είναι σε περίπτωση που αντικαταστήσει τι εθνικέ πρεσβείες πώς η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης θα αντιμετώπιζε εθνικά προβλήματα, ε, διαφορές που έχει ενδεχομένως η Ισπανία με το Γιβραλτάρ, ξέρω εγώ, ή άλλου τέτοιου είδους τύπου ζητήματα. Τέτοιου ζητήματα, μπορείτε να μας το διευκρινίσετε, ευχαριστώ πολύ. Ε, υπάρχει αντιπρόσωπος της Γκου εδώ που θα ήθελε να μιλήσει, όχι... Δίνω λοιπόν στους μη εγγεγραμμένους, ε, στον κύριο Ελζο. Ευχαριστώ. Τρει ερωτήσει έχω για τρία θέματα. Ε, η συνεργασία των μυστικών υπηρεσιών, λέει κύριο Σερενχάουζου. Βεβαίω χρειάζεται να γίνεται αυτή και σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να επεκταθεί. Αλλά παρακαλώ να υπόκειται αυτό σε κοινοβουλευτικό έλεγχο. Και εδώ ανήκει και ο έλεγχο ο δημοσιονομικό. Και σα ερωτώ, τι φρονείτε για την πρόταση να υπάρχει ειδική θέση στον προϋπολογισμό για τις υπηρεσίες αυτές πληροφοριών. Τέλος, ε, δεύτερο μάλλον, διαφάνεια διαβαθμισμένων εγγράφων. Στην έκθεση πεπραγμένων ή δραστηριοτήτων ετησίω δημοσιεύεται, ε, θέλετε να δημοσιεύετε πόσα έγγραφα ε, είναι απόρριτα, είναι διαβαθμισμένα, πόσα έχετε διαβιβάσει, πόσα έχετε λάβει σε άλλε υπηρεσίε. Το έχετε απαντήσει σε ερώτηση αυτό του Κοινοβουλίου. Ε, θα ήταν καλό σε μια τέτοια έκθεση ίσως να δημοσιεύονται αυτά τα στοιχεία. Ε, και ερώτηση τρίτη για τις ε, κατοικίες των υπαλλήλων. Για το 2011 υπολόγισα εκεί τα ποσά. Έχετε υπογράψει συμβόλαια για 66 εκατομμύρια ευρώ. Ξέρω ότι είναι διαφορετική διάρκεια κάθε συμφωλέου ε, ενοικίασης και είναι σχετικό το ποσό αυτό, αλλά θέλω να ρωτήσω το εξή: Το 2012 θα έχουμε αντίστοιχε υπογραφές τέτοιων συμβολέων. Ακούσαμε ότι στο Χονγκ Κόνγκ ε, είναι κατοικία τέτοια και κοστίζει το μήνα 20.000 ευρώ το μίσθωμα. Εκεί τι συμπεριλαμβάνεται, υπάρχουν και ασφαλεία ασφαλείας, είναι μονοτονίκη. Υπάρχει και προσωπικό των επικεφαλής των αντιπροσωπιών που πληρώνεται από αυτό. Και ε, επόμενη ερώτηση. Έχετε εσωτερικές κατευθυντήριες γραμμές για το τι κάνουμε για τις ε, κατοικίες αυτές ε, που μισθώνουμε και μήπως πρέπει το συνολικό κόστος τελικά κάπως να συγκρατηθεί. Ευχαριστώ κύριε Ερενχάουζερ και όλους τους υπολείπους συναδέλφους για την πειθαρχία τους. Θα ήθελα να προσθέσω και εγώ μια μικρή ερώτηση που δεν μπορώ να ρωτήσω τον κύριο Σάλιβαν Ξέρω ότι ως διοικητικός γενικός διευθυντής έχει πολλά καθήκοντα και τώρα έχει αναλάβει και κάποιες περιφέρειες. Ε, κυρία Άστον, είναι τόσο απαραίτητο λοιπόν να τον ε, φορτώνετε τόσο πολύ τον κύριο Σάλιβαν. Πρέπει ο ίδιος να τα όλα αυτά. Μπορείτε να μας απαντήσετε γιατί του έχετε αναθέσει και αυτό το καθήκον, διότι έχει πάρα πολλά άλλα οργανωτικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Γνωρίζω ότι στις 10 και 4 το αργότερο πρέπει να αποχωρήσετε. Ένα τέταρτο νομίζω θα φτάσει. Ελπίζω τουλάχιστον για να απαντήσετε στις ερωτήσεις μου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να μείνω περισσότερο για να απαντήσω όλες τις ερωτήσεις και ευχαριστώ όλα τα μέλη της Επιτροπής για αυτές τις ερωτήσεις. Θα ήθελα κύριε να σας, Γκρέσλα, να σας ευχαριστήσω για όλη σας τη δουλειά. Μιλήσατε για διαφάνεια. Νόμιζα ότι θα μας δίνατε συγχαρητήρια, αλλά ελπίζω να δεχτείτε το γεγονός ότι προσπάθησαν να ξεκινήσω τη σχέση μας με πολύ διαφανή τρόπο. Ευχαριστώ για τα σχόλιά σας όσον αφορά τις προσπάθειες που κάναμε για έξυπνη εξοικονόμηση. Τώρα όσον αφορά τις διαδικασίες πρόσληψης, προσλήψεων. Εμείς προσπαθήσαμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερα μέσω video link, παρότι πολλοί υποψήφοι ε, αισθάνονται ότι δεν τους δίνεται έτσι καλύτερη ευκαιρία, θα προτιμούσαν να είναι εδώ αυτοπροσώπως εγώ λοιπόν όλους τους επιλεγμένους υποψηφίους για επικεφαλής αντιπροσωπείων τους ε, παίρνω συνέντευξη. Προσπαθούμε εάν κάποιος έχει υποβάλει υποψηφιότητα για τρεις ή τέσσερις διαφορετικές θέσεις φροντίζουμε οι συνέντευξεις να λάβουν χώρα την ίδια μέρα. Δηλαδή σε τέτοια περίπτωση θα, δω κάποιον τέτοιο υποψήφιο σε μία μέρα. Και για τις τέσσερις θέσεις είναι απαραίτητο γνωρίζαμε ότι θα έχουμε τεράστιο αριθμό υποψηφίων που θα ήθελαν να συμμετέχουν στην υπηρεσία. Το είχαμε προβλέψει και προσπαθήσαμε να διατηρήσουμε τα κόστη στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο, λαμβάνοντα υπόψη, ωστόσο, ότι οι υποψήφοι για τι θέσει αυτέ προέρχονται από όλο τον κόσμο. Πραγματικά. Μιλάμε για διπλωμάτε, α πούμε. Είχαμε έναν Αυστραλό. Ε, αναπόφευκτα θα, ήταν, θα είχαν έτσι τα πράγματα. Προσπαθήσαμε λοιπόν να είμαστε όσο πιο αυστηροί γίνεται και να αυξήσουμε στο μέγιστο δυνατό το βίντεο, τη βίντεο διάσκεψη ως γενική πρόταση. Σήμερα και πολλές συναντήσεις λαμβάνουν χώρο έτσι, για να ταξιδεύουμε. Το συνολικό ποσό για είναι 28% ε, τα μέλη των κράτων μελών. Είχαμε υποψήφιους πολύ ψηλής ποιότητας. Εγώ θα σας πω ότι ως επικεφαλή αντιπροσωπείας ορίζω τον καλύτερο το καλύτερο άτομο που συνάντησα σε συνέντευξη και εγώ πρέπει να ξέρετε ότι, είμαι, ότι λαμβάνω πίεση από, ομάδες, από λόμπι καθημερινά, άλλες φορές ε, όμορφα, άλλες φορές άσχημα. Προσπαθούμε να λάβουμε ε, να προσλάβουμε υποψήφους από όλα τα κράτη-μέλη, από όλες τις υπηρεσίες. Κάνω ό,τι μπορώ για να έχουμε τους καλύτερους δυνατούς υποψήφιους και για να διορίζουμε τους καλύτερους δυνατούς υποψήφιους και πιστεύω ότι αυτό θα έχει τεράστια σημασία για την φήμη της υπηρεσίας μας. Μιλήσατε για ενημέρωση των κρατομελών. Δεν με εκπλήσει ότι παραπονούνται οι πρέσβεις ότι δεν λαμβάνουν από τα κράτη-μέλη αυτό που πιστεύουν ότι θα έπρεπε να τους παρέχεται. Όλο και περισσότερο ξέρουμε ότι χρησιμοποιούν τα κράτη-μέλη τις πολιτικές μας εκθέσεις. Μπορεί να βάζουν τα δικά τους ε, στοιχεία εκεί και να το στέλνουν πίσω σαν να ήταν δική τους η έκθεση. Εμείς ε, το θεωρούμε αυτό ε, φιλοφρόνηση. Σίγουρα δεν μας πειράζει και ξέρω ότι αληθεύει σε πολλές περιπτώσεις. Υπάρχουν δύο ζητήματα. Το πρώτο είναι ότι Πρέπει να διασφαλίζουμε τη λήψη και την παροχή πληροφοριών ε, αμφίδρομα. Έχουμε και το θέμα της ασφάλειας των πληροφοριών ε, που υποθέτει τεράστια εργασία. Και το δεύτερο είναι η οικοδόμηση της σχέσης με τα κράτη-μέλη ώστε να είναι πολύ πιο άνετη. Το καλά νέα είναι ότι τα πράγματα βελτιώνονται διαρκώς αλλά δεν έχουν φτάσει ακόμα σε άριστο επίπεδο. Κύριε Κάλφιν, με ρωτήσατε χρησιμοποιήσετε ένα, θέλετε ένα παράδειγμα. Εγώ προσπάθησα να χρησιμοποιήσω το παράδειγμα εν μέρη, διότι ο κύριος Ένες μου ζήτησε να δώσω ένα παράδειγμα, αλλά και για να σας ε, δείξω ότι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούμε όλο και περισσότερο με την ΤΕΦΚΟ, για παράδειγμα με τις διάφορες υπηρεσίες, όλο και περισσότερο με τους συναδέλφους από την Κομισιόν, με τους συναδέλφους μου, μελετάμε διάφορες δραστηριότητες. Αναπτύσσουμε λοιπόν μια ε, στάνταρ διαδικασία αν πω λοιπόν στον Επίτροπο, αν μιλάω με τον Επίτροπο Γεωργίας και του μιλάω για δουλειά που κάνουμε σε αγροτικές περιοχές στην αγροτική κοινότητα στην Κίνα, πολύ ενδιαφέρον τομείς και αυτός κάνει τη δική του δουλειά και σε σχέση με αυτό λειτουργεί η δική μας υπηρεσία όταν συνεργαζόμαστε σε θέματα εμπορία. Χθε μιλούσαμε για ζητήματα με τον Μπαγκλαντέ και το τι συμβαίνει εκεί όσον αφορά κάποιε από τι τραγωδίε που έχουν λάβει έχουν συμβεί στον Μπαγκλαντέ, πώς μπορούμε να συνεργαστούμε από άποψη εξωτερική πολιτική και εμπορική πολιτική ώστε να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε τις αλλαγές αυτές τις χώρες. Συνεργαζόμαστε στενά με τους επιτρόπους που ασχολούνται με την απελευθέρωση των θεωρήσεων. Μεγάλο ζήτημα στη δική μα γειτονιά. Αλλά φυσικά να αποκτήσει στο... το Συμβούλιο είναι αυτό που θα λάβει την τελική απόφαση και η Σισίλα Μάλμστρομ έχει ζωτική σημασία σε τι τι ε, συζητήσει και με τον Άντρε Πίλμπαξ ε, στην ΤΕΦΚΟ συχνά συζητάμε για το πώ λειτουργούμε κεντρικά αλλά και πιο σημαντικό τι συμβαίνει επί τόπου. Τα πράγματα δεν είναι τέλεια. Διαρκώ εμφανίζονται νέα προβλήματα. Προσπαθούμε να αναπτύξουμε επίση και μια πλατφόρμα στο πλαίσιο τη οποία θα ασχολούμαστε με ένα σύνολο ζητημάτων ε, συζητώντα με όλου. Αυτό προεδρεύεται συχνά από μένα, άλλε φορέ τον Πιέρ Εκεί θέλουμε να συμμετέχουν όλε οι υπηρεσίε που σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο τομέα. Η Συρία, για παράδειγμα, είναι ένα, κάτι που συζητάμε τακτικά, το Μάλι. Εκεί θέλουμε να συμμετέχουν όλοι όσοι μπορούν να συνεισφέρουν σε, στη συζήτηση αυτή. Προσπαθούμε λοιπόν να επιτύχουμε τον καλύτερο δυνατό συντονισμό. Σε ορισμένε περιπτώσει έχουμε συγκεκριμένα στάνταρ, μια τυπική διαδικασία. Σε άλλε περιπτώσει όπως όταν συζητούσαμε με τη Μαρία Δαμανάκη για τα αλληλευτικά ζητήματα ή με άλλους για τη Σομαλία, όλες οι συνέργειες που μπορούμε να κάνουμε βελτιώνονται, δεν είναι ακόμα τέλειες. Τώρα, όσον αφορά την απόσπαση προσωπικού των κρατών μελών, έχουμε δύο ίδια ανθρώπων, διπλωμάτες που έρχονται στην υπηρεσία για έως και 10 χρόνια. Αυτοί πληρώνονται από εμάς, δεν κοστίζουν τίποτα στο κράτος μέλος. Κατά καιρούς ε, Έχουμε απεσπασμένου εθνικού εμπειρογνώμονε από τα κράτη-μέλη, για του οποίου πληρώνουν τα κράτη-μέλη, αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι με του οποίου συνεργαζόμαστε εμεί, που προέρχονται από τα κράτη-μέλη, του απασχολούμε εμεί, του πληρώνουμε εμεί. Συνεπώ αυτό δεν αποτελεί ζήτημα σίγουρα. Τα κράτη-μέλη που αυτή τη στιγμή εφαρμόζουν λιτότητα στι ε, ομάδε του σε όλο τον κόσμο, ε, Μα στέλνουν ε, ε, ανθρώπους υψηλή ποιότητας ε, να εργαστούν στην υπηρεσία. Όσον αφορά την καλύτερη χρήση των εθνικών πόρων, Μόλι έχει ξεκινήσει η υπηρεσία, προσπαθούμε να συνεργαζόμαστε όλο και περισσότερο με τα κράτη-μέλη και να τα πείθουμε να συνεργαζόνται όλο και περισσότερο με εμά. Με ορισμένα κράτη-μέλη εργαζόμαστε καλύτερα, με άλλα λιγότερο. Κάποιοι βασίζονται σε εμά γιατί είναι μικρότερα κράτη και εξαρτώνται από μας. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι συνεργασίας με τις εθνικές υπηρεσίες. Βελτιώνονται διαρκώς. Αλλά φυσικά, ναι, τα πράγματα δεν έχουν φτάσει σε κάποιο άριστο επίπεδο ακόμα. Για να απαντήσω τώρα στον κύριο Σκυλακέκη. Οι διαδικασίες διαπραγμάτευσης για ε, διαγωνισμούς ε, ε, προμηθειών είναι δύσκολο. Δεν έχουμε αρκετού προμηθευτέ ώστε να εφαρμόσουμε επαρκεί διαδικασίε διαγωνισμών. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για τα 60.000 ευρώ, όπω είπατε, που είναι σημαντικά χρήματα, να εφαρμόζουμε διαγωνισμού όπου μπορούμε. Ε, ακριβώς για τους λόγους του οποίους αναφέρατε με ρωτήσατε για του κατοικίε στο Χονγκ Κόνγκ στη Τζαμαϊκά ε, πρέπει να δείτε το πώ είναι το τοπίο στην κάθε χώρα ε, στο Χονγκ Κόνγκ έχετε τεράστιου ουρανοξύστες με μικρά διαμερίσματα, ενώ στη Τζαμάικα τα σπίτια είναι συνήθω μεγαλύτερα. Έχουμε προβλήματα με κάποιες από τις κατοικίες. Εγώ είχα ζητήσει μία αξιολόγηση κάθε ε, επιμέρους κατοικίας που έχουμε, διότι ορισμένε από αυτές χρειάζονται μεγάλες επισκευές, ε, είναι κακές συνθήκες διαβίωσης και αλλού έχουμε λάβει κατοικίες οι οποίες θα μπορούσαν ίσως να χρησιμοποιηθούν καλύτερα, να αξιοποιηθούν καλύτερα και σε ορισμένα άλλα μέρη έχουμε κατοικίες που χρησιμοποιούνται επίσης και για πολλές από τις συνεδριάσεις των αντιπροσωπιών. Πρέπει να καταλάβετε ότι σε τέτοιες μεγάλες κατοικίες υπάρχουν και πολλά γραφεία μέσα στο ίδιο κτίριο σε πολλές χώρες το 20-30% της κατοικίας χρησιμοποιείται ως γραφειακός χώρος διότι τα γραφεία δεν είναι αρκετά μεγάλα. Έτσι λοιπόν τα κτίρια είναι μεγαλύτερα γιατί χρησιμοποιούνται διαφορετικά σε άλλα μέρη. Οι κατοικίες είναι απλά κατοικίες. Ε, οπότε πρέπει να γνωρίζει κανείς ε, τι ακριβώς συμβαίνει σε κάθε χώρα ώστε να μπορεί να αξιολογήσει κατά πόσο έχουμε τη σωστή ποιότητα κατοικίας για να μπορέσει κάποιος να ζήσει, να δεχθεί κόσμο, δεν χρειάζεται αίθουσα υποδοχή, είναι κομμάτι της δουλειά και να υπάρχει και αρκετό χώρο γραφείων για όλου. Και εμεί έχουμε προβλήματα σε ορισμένε περιοχέ. Για πολλά χρόνια, 40 χρόνια μερικέ φορέ, είχαμε νοικιάσει κάτι, ενώ θα έπρεπε να ήταν προτιμότερο να είχαμε αγοράσει πριν από 25 χρόνια και να είχαμε εξοικονομήσει πολλά χρήματα. Με βάση του νέου κανονισμού λοιπόν θα μπορέσουμε να λειτουργήσουμε πιο δημιουργικά και να μην ξοδεύουμε, να μην σπαταλάμε χρήματα όταν σε ένα μέρος είναι προτιμότερο να αγοράσουμε αντί να νοικιάσουμε άλλα. Όταν βλέπετε τα τραγωνικά μην νομίζετε ότι μιλάμε για ανάκτορο, δεν είναι απαραίτητα ανάκτορο. Σε ορισμένα μέρη φαίνεται να είναι πολύ ωραίο, αλλά δεν θα έλεγα ανάκτορο, ε, ειδικότερα σε σύγκριση με ε, τα κτίρια πρεσβείων. Μας ρωτήσατε κατά πόσο θα μπορούσαμε να έχουμε ένα ανεξάρτητο φάσμα επιθεωρητή, συγγνώμη. Έχουμε ε, άνθρωποι που πηγαίνουν, πηγαίνουν και αξιολογούν τι γίνεται στις διάφορες αντιπροσωπείες. Είναι και μια υπηρεσία υποστήριξης, εξετάζει τη λειτουργία της διοίκησης, την αποτελεσματικότητα, την ποιότητα διαβίωσης των ατόμων, την ασφάλεια, τον τρόπο αποτελεσματικής συνεργασίας των ατόμων, διότι έχουμε άτομα που συνεργάζονται από διαφορετικές χώρες, διαφορετικά θεσμικά όργανα και τους ζητάμε να συνεργαστούν αποτελεσματικά. Λειτουργεί πολύ καλά, αλλά αυτή η υπηρεσία μπορεί να μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε και διάφορα προβλήματα, ζητήματα και να παρέχουμε και συμβουλές για καλύτερες μεθόδους, καλύτερη χρήση περαιτέρω κατάρτιση, ενδεχομένως οικονομικά θέματα του προσωπικού, διότι η κατάρτιση θα βοηθήσει στην ανάπτυξη ταυτότητας της υπηρεσίας. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό θα μπορέσει να διασκεδάσει τις ανησυχίες σας για αυτά που αναφέρατε. Ε, μου αναφέρατε για την δημοσιονομική ουδερεότητα. Όταν εμείς αναλάβαμε την υπηρεσία, θέλαμε αυτό το αμάλγαμα που δημιουργούμε να μην κοστίζει περισσότερο από ό,τι κόστιζε προηγουμένως. Έτσι εννοούσαμε ουδέτερα. Με αυτό ενώσαμε όταν είπαμε ουδετερότητα. Όταν στην αρχή ωστόσο δεν λάβαμε τους απαραίτητους πόρους και ζητήσαμε διόρθωση αυτού. Δεν έχω λοιπόν αναθετήσει την υποσχέσή μου. Και ευχαριστώ που μου δίνετε δυνατότητα να το τονίσω διότι στις παρούσες οικονομικές συνθήκες πρέπει οπωσδήποτε να είμαστε φιδωλοί. Έχουμε ε, ε οδηπορικά, κόστος ταξιδιού, είπα χρησιμοποιούμε συνδέσεις βίντεο όπου μπορούμε έχουμε περικόψει τα μέλη των αντιπροσωπιών που ταξιδεύουν ανά πάσα στιγμή προσπαθούμε να είμαστε βέβαιοι ότι όταν μας επισκέπτεται κόσμος από διάφορα μέρη του κόσμου για εκπαίδευση και ούτω καθεξής ότι αξιοποιούμε στο μέγιστο δυνατό τις ημέρες που περνούν μαζί μας και προσπαθούμε να κόψουμε, ε, να περιορίσουμε οποιοδήποτε κόστος, αλλά όπως καταλαβαίνετε το μεγαλύτερο σταθερό κόστος, γενικό κόστος είναι το προσωπικό. Μας έχει δοθεί τεράστιος αριθμός προσωπικού, αυτός είναι ο αριθμός που έχουμε, δεν μπορούμε να του στείλουμε πίσω και συνεπώς πρέπει να τους πληρώσουμε και να τους ταΐσουμε. Και αυτό σημαίνει ότι κληρονομώ εγώ όλα τα ζητήματα που αφορούν τις, ε, ε, ε τους προβασμούς των ατόμων, τις προαγωγές των ατόμων και όλα τα σχετικά ζητήματα. Εγώ νομικά υποχρεωμαι να δώσω στον κόσμο ό,τι δικαιούται. Και αυτό είναι κομμάτι των των πόρων, διότι δεν μιλάμε εδώ ότι δημιουργήσαμε νέα χρήματα στο σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι αυτός ο κόσμος δεν θα βρισκόταν μαζί μας. Τώρα όπως είπατε σε περίπτωση όπως το Αφγανιστάν στη Μογκαντήσο είναι σημαντικό να ε, ε, δώσουμε στους ανθρώπους κάποια ανταμοιβή ε, όταν τους έχουμε βάλει να εργαστούν σε ένα τόσο δύσκολο περιβάλλον. Πραγματικά έχουμε εντυπωσιασμένοι από το εκπληκτικό έργο όλων αυτών των ατόμων για λογαριασμό μας. Είναι από τις πιο δύσκολες συνθήκες που θα μπορούσε να φανταστεί κανείς. Ζητήσαμε από το επικεφαλής αντιπροσωπιών από το Προεδρείο των αντιπροσωπιών να εξετάσει αυτά τα ζητήματα των ε, ημερών διακοπών και όλα αυτά διότι όπως είπα και εγώ θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι καλύτερο το είπαν και αυτοί το θέμα είναι ότι δεν μπορώ να προτείνω αλλαγές η πρόταση πρέπει να προερθεί από την Κομισιόν και όπως γνωρίζετε αυτή τη στιγμή ε, ασχολούνται με μια μακροχρόνια άσκηση για πολλά θέματα, αλλά θέλουμε να του ζητήσουμε διότι χρειάζεται κάποια αλλαγή στον κανονισμό. Τα πράγματα οριμάζουν κάποια στιγμή και χρειάζεται να τα αναθεωρήσουμε. Αλλά οι αντιπροσωπείε γνωρίζουν πολύ καλά ότι πρέπει να εξετάσουμε το ζήτημα πολύ προσεκτικά. Δεν νομίζω ότι έχουμε τεράστια γραφειοκρατία ε, και θεσμική και έχει και όλα αυτά που είπατε. Πιστεύω ότι σίγουρα έχουμε κάποιες δυσκολίες επειδή βρισκόμαστε στα αρχικά στάδια. Φέρνουμε κόσμο από διαφορετικά θεσμικά όργανα στο ίδιο κτίριο. Αυτό προϋποθέτει κάποιες δυσκολίες. Αλλά υπάρχει μια αίσθηση ομάδας και ε, Πολλοί έχουν εγκαταλείψει συναδέλφου με του οποίου συνεργάζονταν σε άλλα κτίρια και φυσικά υπήρξε κάποια αβεβαιότητα. Έπρεπε να επανατοποθετήσουμε τον καθένα, να φροντίσουμε ο καθένα να έχει μια θέση, καθήκοντα, να έχει δυνατότητε για το μέλλον. Πιστεύω λοιπόν ότι φέτο όλα τα πράγματα αυτά θα ομαλοποιηθούν, αλλά τα πράγματα ήταν δύσκολα. Δεν υπάρχει αμφιβολία και ειδικά όταν έχουμε πολλού διπλωμάτε που έρχονται από διάφορα κράτη-μέλη. Ναι, η ζωή δεν είναι αυτή έχει αλλάξει για πολλά, πολλούς από αυτούς τους ανθρώπους τώρα όσον αφορά τη δημοσιονομική στήριξη. Συμφωνώ ε, και με εσάς και με το ελεκτικό συνέδριο πρέπει να το εξετάσουμε προσεκτικό και αναφέρατε κάποια ενδιαφέροντα παραδείγματα. Εγώ αναφέρω όμως σε παραδείγματα όπως ε, το Αφγανιστάν όπου υπάρχουν όλα τα ζητήματα που γνωρίζουμε τόσο καλά για το πώς πρέπει τελικά να αναπτυχθεί αυτή η χώρα πρέπει να αναπτύξει και τις δικές της δυνατότητες. Αυτό αληθεύει για πολλές χώρε σε όλο τον κόσμο. Το ζήτημα λοιπόν είναι να βρούμε τρόπους στήριξης της ανάπτυξης των κρατικών συστημάτων με τρόπο τέτοιο που εμείς αναγνωρίζουμε ως διαφανή και σωστό και που να επιδέχεται οικονομικό έλεγχο θα πρέπει να τους δώσουμε υπευθυνότητα, να τους αναθέσουμε υπευθυνότητα στους ίδιους, πρέπει να το κάνουν μόνοι τους. Αυτό φυσικά δεν πρέπει να γίνεται εις βάρος ε, της διασφάλισης ε, της σωστής ε, χρήσης των ε, ευρώ των φορολογουμένων. Δεν μιλάμε για αύξηση του προϋπολογισμού κατά 500 εκατομμύρια. Το βλέπετε λάθος. Ήταν χρήματα που υπήρχαν στο παλιό σύστημα. Δεν αυξήσαμε τον προϋπολογισμό για τη δημιουργία τη υπηρεσία. Όταν μίλησα για μεγαλύτερη δέσμευση στη Μέση Ανατολή, θα μπορούσα να σας πω, μιλήσω πιο λεπτομερώς για πολλά πράγματα, για τα οποία η παρουσία της ΕΕΔ κάνει μεγάλη διαφορά. Αλλά η ερώτηση που μου κάνατε είναι κατά πόσο θα αντικαταστήσουμε τις εθνικές πρεσβείες. Όχι, δεν είμαστε κράτος μέλος, δεν κάνουμε ό,τι κάνουν τα κράτη-μέλη. Κάνουμε αυτό που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είτε πρόκειται για συντονισμένη προσέγγιση κοινή εξωτερικής πολιτικής, ε, οι απόψει που παγιώνουμε μέσω συμπερασμάτων του Συμβουλίου, η εργασία που κάνουμε στην Κομισιόν και στο Κοινοβούλιο για θέματα εμπορίου, κλιματικής αναλλαγή ως το πώς υποστηρίζουμε αναπτυσσόμενες χώρες, ε, διαχείριση κρίσεων, όλα αυτά. Όλα αυτά κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που ε, από τις δραστηριότητες των κρατών μελών. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι χώρε, ε, όπως η Ισπανία για παράδειγμα, δεν θέλουν να στείλουν διπλωμάτες τους στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική δράση, Ας πούμε, όταν ε, θέλουν να εξορθολογήσουν την ύπαρξη πρεσβειών οι χώρες τους, ε, για παράδειγμα. Θα μπορούσαμε δηλαδή να μιλήσουμε για κάποιο είδου ευρωπαϊκή πρεσβεία όπου θα συμμετείχαν μια σειρά κρατών μελών και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση και θα λειτουργούσαν μαζί και αυτό θα μπορούσε να μα μειώσει τα κόστη και να χρησιμοποιήσουμε πιο αποτελεσματικά του πόρου. Έχουμε λοιπόν συμφωνίε με κάποια κράτη-μέλη για κάτι τέτοιο κάποια στιγμή σε ορισμένα μέρη. Επίση έχουμε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων που συστεγάζεται μαζί μα σε ορισμένα μέρη του κόσμου και με άλλε υπηρεσίε. Το κάνουμε δηλαδή αυτό, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα κλείσουμε πρεσβείε. Δεν σημαίνει ότι θα κάνουμε τη δουλειά των κρατών μελών. Μου ζητήσατε επίσης, ε, με ρωτήσατε επίση όσον αφορά τα διαβαθμισμένα έγγραφα και τη συνεργασία πληροφοριών. Δεν ξέρω τι εννοείται διαβαθμισμένα έγγραφα που πέρασαν από ποιον σε ποιον. Εμεί έχουμε τη δυνατότητα να μπορούμε να αντλήσουμε πληροφορίε που θέλουν να μα δώσουν τα κράτη-μέλη ώστε να μπορούμε να έχουμε κάποιε πληροφορίε και να κατανοούμε καλύτερα τι συμβαίνει σε ένα συγκεκριμένο μέρο του κόσμου. Είμαστε τυχεροί που κατά καιρού στην υπηρεσία μας καταφέραμε να πάρουμε πληροφορίες που μας παρήχαν και οι υπηρεσίες πληροφοριών. Τα έγγραφα που έρχονται σε μένα έχουν γραφτεί για εμένα και έρχονται για αυτό το σκοπό. Είναι πληροφορίες διαθέσιμες για τα ανώτερα στελέχη τους Προέδρους του Συμβουλίου και της Κομισιόν, πληροφορίες που πηγαίνουν προς επιτρόπους ανάλογα με το θέμα. Είναι δύσκολο λοιπόν να σα απαντήσω αυτή την ερώτηση, να σα πω τι πηγαίνει πού, διότι έχουμε τεράστια ροή πληροφοριών διαρκώ. Βασιζόμαστε σε τεράστιο βαθμό στι ερχόμενε και εξερχόμενε πληροφορίε από τα κράτη-μέλη, από τι αντιπροσωπείε μα, από ανοιχτέ πηγέ, από το γεγονό ότι έχουμε μια υπηρεσία που λειτουργεί 24 ώρε το 24ωρο, στι εισερχόμενε ημέρε τη βδομάδα, παρακολουθώντα τι αντιπροσωπειε μα απο ανοιχτε πηγε απο το γεγονο οτι εχουμε μια υπηρεσια που λειτουργει 24 ωρε το 24 ωρο 7 ημερε τη εβδομάδα παρακολουθωντα τι συμβαινει στον κόσμο μέσω ραδιοφωνικών τηλεοπτικών καναλιών, αντιπροσωπείων κ.ο.κ. Όσον αφορά τη στελέχωση, αυτά που εξήγησα για το, η διαφορά μεταξύ Χονγκ και Τζαμάικας, με τις αυξομοιώσει του ευρώ το κόστος διαφέρει. Εάν ε, σε κάποιε περιπτώσεις αν ε, χάσει αξία το ευρώ σε σχέση με κάποιο νόμισμα τότε τα πράγματα κοστίζουν περισσότερο. Προσπαθούμε να κάνουμε ορθολογική χρήση των πόρων ειδικότερα όσον αφορά τις κατοικίες. Ε, αναφέρθηκα επαρκώς νομίζω σε αυτό το ζήτημα. Και τώρα όσον αφορά τον ορισμό ανώτατων ορίων, προσπαθούμε στο μέγιστο βαθμό να διασφαλίσουμε ότι δεν ξοδεύουμε παραπάνω από ό,τι έχουμε στη δυνατότητά μας. Δεν προσπαθούμε να παρέχουμε ανάκτορα, προσπαθούμε να παρέχουμε μια επαρκή κατοικία σε κάποιον, αλλά πρέπει να καταλάβετε ότι στο Χονγκ για παράδειγμα, αν προσπαθεί κανεί να αγοράσει ή να νοικιάσει, αυτό κοστίζει πολύ περισσότερο από την ενοικίαση ε, ίδιο τύπου ιδιοκτησία σε άλλο μέρος του κόσμου. Και τέλος κύριε Πρόεδρε, ο Ντέβιτ Σάλιβαν κάνει καταπληκτική δουλειά στο ρόλο που του έχω αναθέσει, τον οποίο γνωρίζετε. Το να διασφαλίζει ότι όλη η επιχείρηση αυτού του οργανισμού, όχι μόνο στα κεντρικά αλλά και σε όλο τον κόσμο, η διοίκηση, η οικονομική διοίκηση και όλα αυτά, να αναφέρεται απευθείας σε αυτόν. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε το τεράστιο ταλέντο που κάθεται δίπλα μου. Το γνωρίζαμε όταν ήταν στην Γενική Διεύθυνση Εμπορίου. Έχει τεράστια εμπειρία και είναι και φυσικά και διπλωμάτης. Με τον Πιερ λοιπόν τον κάλεσα να δει τον πλανήτη και να πει, να δει πού θα μπορούσαν να συνεργαστούν μαζί. Ο οποίος, λοιπόν ενδιαφέρεται ιδιαίτερα στη σχέση μας με την Κίνα όπου τα εμπορικά και οικονομικά ζητήματα είναι τεράστια σημασία. Ενδιαφέρεται ιδιαίτερα στη σχέση μας με τη Ρωσία, όπου και πάλι είναι πολύ σημαντικά αυτά τα ζητήματα. Προσπαθούμε δηλαδή να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο βαθμό του πόρου μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Yeah, thank you very much for Εμείς σας ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος μια που μας εφηρώσατε τόσο χρόνο για να απαντήσετε στις ερωτήσεις μας και γνωρίζουμε ότι τώρα θα πρέπει να προλάβετε το αεροπλάνο για να πάτε στην Ιρλανδία επευκαιρία ευκαιρία της Προεδρίας της χώρας και σας ευχαριστούμε όχι μόνο που ήρθατε εδώ και απαντήσετε τις ερωτήσεις αλλά ε, πρέπει να σας ευχαριστήσουμε ε, νομίζω ήρθε η ώρα για όσο επιτελείται για την Ευρωπαϊκή Ένωση γενικά οπότε ε, σας ευχόμεθα καλή τύχη, καλή επιτυχία και φέτος. Um, λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, ο κύριος Σάλιβαν ε, θα απαντήσει στο δεύτερο γύρο των ερωτήσεων, ε, προσεφέρθη ευγενικός και ε, παρακαλώ να αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία. Ο Ζαμπιεροντή θέλει πρώτο το λόγο και μετά η κυρία Γιάλα. Σαλαφράγκα, Γκρέσλε και λοιποί. Άρχεται λοιπόν η συζήτηση. Ζαμπιεροντή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η κατάσταση είναι όλο ιδιάζουσα. Εκφράζω τη λύπη μου που δεν είχαμε αυτή την ανταλλαγή απόψεων πέρυσι, διότι η υπηρεσία συστάθηκε την 1η Δεκεμβρίου του 2009 από τη συνθήκη της Λισαβόνας, ακόμα και αν χρειάστηκε χρόνο να εγκατασταθεί. Η απόφαση είναι το 2010. ξέρω, στο λειτουργικό πλαίσιο είναι μόλις το 2011 και το επιχειρησιακό, αλλά λυπάμαι που για το 2010 δεν είχαμε αντίστοιχη ανταλλαγή απόψεων για να προετοιμάσουμε ε, δεόντως τις συζητήσεις μας. Κρίμα λοιπόν που δεν κάναμε αυτή τη συζήτηση και πέρσι. Γνωρίζετε Πρόεδρε ότι έχω μεγάλη επιφύλαξη για αυτές τις επιμέρους απαλλαγές που δίνει η Επιτροπή μας στις διάφορες υπηρεσίες. Απορρίψαμε ε, την απαλλαγή την αρνηθήκαμε για το Συμβούλιο χωρίς καμία πολιτική συνέπεια, πάντες το ξέχασαν. Ε, εγώ και για την Κομισιόν το ίδιο έγινε, διαιρωτώ με. Ποια απαλλαγή θα δώσουμε τώρα σε αυτά τα επιμέρους όργανα. Και θα ήθελα να σας ε, παρακαλέσω, Πρόεδρε, να μας ενημερώσετε ε, ποιος είναι ο περίμετρος του λογιστικού ελέγχου. Δηλαδή, επί ποιου θα δώσουμε εμείς απαλλαγή Ποια είναι λοιπόν η περίμετρος ε, των διοικητικών και των ε, επιχειρησιακών και των λειτουργικών δαπανών. Ο κύριος Φίλε, ο κύριος Πίμπαλξ, ε, ποιοι είναι οι αρμόδιοι επίτροποι. Σε ποιον λοιπόν χορηγούμε απαλλαγή και για ποιες δράσεις. Τρία είναι τα μέλη του ελεγκτικού συνεδρίου που ελέγχουν το σύνολο αυτών των δραστηριοτήτων, αλλά ξαναρωτάω ποια είναι η περίμετρος, ε, σε τι πράγμα εμείς δίνουμε απαραγή, πολιτικά. Και ένα σχόλιο έχω, μια παρατήρηση. Εδώ και ένα χρόνο ζητώ να κάνουμε ένα λογιστικό έλεγχο για τις οικονομίες που θα μπορούσαμε να κάνουμε σε συνεργασία σε τρία επίπεδα δημοσίων δαπανών, Ευρώπη, κράτος, περιφέρεια. Υπάρχουν τομείς, ας πούμε, η έρευνα, η διεθνής μας παρέμβαση, η παρουσία και η διπλωματία. Μπορούμε να κάνουμε οικονομίες από μια συντονισμένη δράση. Δεν έχει έρθει η ώρα να έχουμε μια πολιτική αξιολόγηση των δράσεων που κάνουμε ε, στα κράτη-μέλη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έναν ανεξάρτητο λογιστικό έλεγχο που θα μπορούσε να κάνει το ελεγκτικό συνέδριο, το ευρωπαϊκό σε συνεργασία με τα 27 εθνικά ελεγκτικά συνέδρια. Με μετάφραση στις γλώσσες μας για να συζητήσουν τα ευρωπαϊκά και τα εθνικά κοινοβούλια για να δούμε πώς θα κάνουμε οικονομίες. Έχουμε εκατοντάδες κτίρια κάθε φορά που πάμε στο εξωτερικό ε, το συνειδητοποιούμε. Οι πρεσβείες και οι υπηρεσίες δεν μοιράζονται ούτε ένα φωτοτυπικό μηχάνημα. Καλά τώρα τα παραλέω, αλλά κάθε φορά που ταξιδεύουμε αυτή την αίσθηση αποκομίζουμε. Εντάξει, ε, βρίσκονται δίπλα-δίπλα στις ε, συσκέψεις που κάνουν εργασίας, αλλά μπορούμε να κάνουμε μία απογραφή ε, των ε, εξοικονομήσεων που θα μπορούσαμε να κάνουμε αν συνεργαζόταν οι πρεσβείες, οι διπλωματίες των κρατών μελών και η νεότευκτη δική μας υπηρεσία. Τελευταία ερώτηση. το κείμενο που μας δόθηκε είναι μόνο στα αγγλικά. Μήπως θα μπορούσατε να το μεταφράσετε στις 4-5 γλώσσες για να ενημερωθούμε. Ευχαριστώ. Η κυρία Γιάλα Σέντερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ να ευχαριστήσω την ε, πάντια εκπρόσωπο. Ήταν πάρα πολύ χρήσιμο όσο ακούσαμε, ε, ε, Πώ είναι η κατάσταση, πόσο δύσκολα είναι αυτή η τεχνογνωσία, το know-how που έχουμε και σε σχέση με τον κύριο ο Σάλιβαν, συμφωνώ με τα όσα μας εξηγήθηκαν. Επομένως, να δούμε σε σχέση με το παρελθόν τι μπορούμε να αλλάξουμε για το μέλλον για την αντιμετώπιση των κρίσεων και με αυτά τα οποία ακούσαμε είμαι σίγουρος ότι η ΕΙΕΔ θα αποσπάσει και άλλα βραβεία όπως ε, τα βραβεία που πήρε η Ευρωπαϊκή Ένωση πέρσι. Υπάρχει πολιτική βούληση. Όλα αυτά επομένως να ευοδοθούν. Τώρα έχω κάποιες ερωτησούλες. Πρώτα πρώτα σε σχέση με την κινητικότητα. Σε κάποιες περιπτώσεις ερωτώ η γενική διπλωματία διακρίνεται από κινητικότητα. Η κινητικότητα τέλο πάντων των διπλωματιών των εθνικών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάπω διαφορετική, η Κομισιόν έχει άλλες ανάγκες, ε, κάποια διοικητικά θέματα και όσον αφορά τις αντιπροσωπείες σας ερωτώ τι είδου κινητικότητα θα ισχύσει, διότι σε κάποιες περιπτώσεις, όπως είπαμε, υπάρχουν ε, θέματα των υπηρεσιών πληροφοριών, ε, το, το know-how αυτής της νέας διπλωματίας, Οπότε θα πρέπει η κινητικότητα να μην είναι ένα εμπόδιο σε κάποιες διαδικασίες εκπαίδευσης, προσαρμογής. Και η κινητικότητα βέβαια εξορισμού θα πρέπει να μην είναι να είναι αναπόσπαστο τμήμα των όσων κάνει μια αντιπροσωπεία. Ε, μετά, σε σχέση με τα όσα έλεγε για την συνεργασία ο κύριος Σοντή και για μας, ε, την Ισπανία, ο Υπουργός ε, Μαργάγιο επίσης κάνει μια τέτοια προσπάθεια γιατί καμιά φορά η κρίση προσφέρει κάποιες ευκαιρίες προς εκείνη την κατεύθυνση δηλαδή να δούμε πώς θα μπορέσουμε τελικά να έχουμε συνεργασία στην πλωτικό επίπεδο στην Ευρώπη. Και να δούμε κατά πόσο συμφωνούν τα κράτη-μέλη με το να έχουν συνεργασία, ούτω ώστε να μην έχουμε επικαλύψεις ενεργειών. Επίσης, για πέστε μας, τι γίνεται με το προσωπικό, με, με αυτούς οι οποίοι τέλο πάντων επαναπατρίζονται από κάποιες ε, περιπτώσεις ε, κατεπιούσης ανάγκης, όπως ε, αυτοί που επαναπατρίστηκαν από την Συρία. Φυσικά και θα εξυπηρετούσαν να μένανε εκεί, αλλά ήταν η ασφάλειά τους που διακυβευόταν. Επομένως, τι γίνεται. Τι τους κάνουμε εδώ μέχρι ότου πάνε ξανά κάπου αλλού. Και τώρα για τον κύριο Κάρελ Πίνστεν, αφού τον ευχαριστήσουμε για το έργο που έχει επιτελέσει τόσο νεωτερικό και καινοτόμο, τι διαφορετικά προβλήματα έχουμε στην ΕΕΔ σε σχέση με τα προβλήματα που συνήθως αντιμετωπίζονται σε άλλα θεσμικά όργανα. Έχουμε κάτι το διαφοροποιημένο ή απλώς για άλλη μια φορά αντιμετωπίζουμε τα διοικητικά Αυτά που γίνονται συνήθως στους οργανισμούς όπου τέλος υπάρχουν ε, τέτοιες λειτουργίες και συμβάσεις. Αφγανιστάν, Σαχέλ, ε, σε αυτά τα μέτωπα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Αγιάλα, Ο κύριος Σαλαφράγκα, επόμενος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Πρώτα-πρώτα θα πρέπει να ευχαριστήσουμε την ε, Λέδη Άστον για τα όσα μας, μας εξήγησε και για το ότι απάντησε αυτές τις 140 τόσες ερωτήσεις. Mm. Δεν, νομίζω ότι είναι κάπως λαϊκιστικό το να ασχολούμεθα με το πόσα τετραγωνικά μέτρα είναι το, το γραφείο, ο χώρος τέλος πάντων του επικεφαλής της κάθε προσωπίας. Βεβαίως θα πρέπει να έχουμε συμπληρωματικότητα, να, να, να άρουμε κάποιες δυσλειτουργίες, να προβάλλουμε περισσότερο την Ευρωπαϊκή Ένωση και να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Πολύ σημαντικό αυτό. Το σούτο μάλλον καθότι περνάμε περίοδο κρίσης. Άρα θα πρέπει να ενεργήσουμε έτσι ε, σε πνεύμα λιτότητος και υπευθυνότητος. Στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων υπονοούμε μια έκθεση σχετική σε αυτό το πνεύμα. Οπότε είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη ότι αυτή είναι η πρώτη προσπάθεια που γίνεται για να αναλύσουμε έτσι τη διαδικασία της απαλλαγή και άρα να μην ξεχνούμε τα όσα μας έχει πει το ελληνικό συνέδριο. Ότι δηλαδή δεν είχαμε τίποτα σοβαρά σφάλματα όσον αφορά τις ε, δαπάνες Άρα είπαμε να έχουμε πνεύμα λιτότητος, αλλά όχι υπερβολές. Γιατί ακριβώς δεν θα πρέπει μέσω της ε, απαλλαγής να υπονομεύσουμε κάποια βασικά στοιχεία, κάποιες αποφάσεις τελικά που λαμβάνονται και που διέπουν την ΑΕΔ. Πρέπει να εφαρμόζεται με προσοχή η νομοθεσία όσον αφορά τις ε, συμβάσεις πρόσληψης. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το τι διέπει την κάθε σύμβαση, την κάθε πρόσληψη, τι προβλέπεται κάθε φορά. Άρα, θα πρέπει να προσέξουμε και τις αποστολές παρατήρησης εκλογών, που είναι κάτι που μπλέκεται άμεσα στο κοινοβούλιο. Άρα, πάντα λέμε ναι σε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες και θα πρέπει να δούμε επίσης τι γίνεται όσον αφορά τους υψηλόβαθμους υπαλλήλους και τι γίνεται όσον αφορά τους, τους χαμηλόβαθμους, τι ποσοστά ε, συντρέχουν εδώ, τι γίνεται με τη, με τη χρησιμοποίηση ε, στρατιωτών στις αποστολές εκείνες. Να δούμε επίσης σε ποιο βαθμό χρησιμοποιούμε την ανάλυση κόστου ωφέλους ποιες ε, αντιπροσωπείες δεν αποδίδουν και δεν θα έπρεπε να είναι ανοιχτέ. Πού υπάρχει υποστήριξη, πλαισίωση, σε, σε ποιες χώρες. Οπότε θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα όσα συζητούνται στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και συμφωνώ με την κυρία Άστον, τη Λέδη Άστον, όσον αφορά τις αρμοδιότητες και ικανότητες του κύριου Αουσάλιβεν, τον οποίο και γνωρίζω περισσότερο από 30 χρόνια. Ευχαριστώ κύριε Σαλαφαρανκά. Θα ήθελα να αξιοποιήσω την ευκαιρία εξ ονόματος Επιτροπής μας για να πω ότι για μας είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η συνεργασία με τις επιμέρους επιτροπές και εξού και οι ε, προτάσεις, οι απαιτήσει της ΑΦΕΤ ε, τις οποίες ακολουθούμε. Η απαλλαγή δεν αφορά αποκλειστικά τη δική μας Επιτροπή, την Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού, αλλά τα ε, γενικότερα συμφέροντα του Κοινοβούλιο. Εξού και το Κοινοβούλιο εγκρίνει ή απορρίπτει την απαλλαγή και είναι σημαντικό να συνεργάζονται όλες οι επιτροπές. Ευχαριστώ κύριε Σαλαφράκα και για την γνωμοδότηση εξ τη Επιτροπή Εξωτερικών. Η κυρία Γκρέσλε είναι η επόμενη στον κατάλογο μου. Ευχαριστώ. Κύριο Σάλιβαν, δυστυχώ εσά πέφτει ο κλήρο τώρα και θα επιμείνω γιατί δεν μου απαντήθηκαν από την ύπατη εκπρόσωπο κάποια πράγματα. Πρώτον, σα είπα ότι επιλεκτικά δρούν τα κράτη-μέλη στι θέσει. 40% των πρέσβεων είναι πρέσβει από τα κράτη-μέλη. Είχαμε συνεννοηθεί για ένα τρίτο ε, και μάλιστα εγκάρσια, όχι μόνο τα ανώτατα στελέχη, γιατί αυτό το ένα τρίτο έγινε 40%. Ότι παίρνετε πάντα τους καλύτερους, συγγνώμη, αλλά μου δημιουργεί αυτό μηδίαμα. Κοίταξα πώς είναι οι διαδικασίες προσλήψεων και από αυτά που ακούω ξέρω ότι σε πολλές περιπτώσεις είναι φωτογραφικές οι διατάξεις. Ξέρουμε από την αρχή ποιο θα πάρουμε. Και ορισμένοι δηλώνουν υποψηφοί ότι δεν πρόκειται να συμμετέχουν σε άλλη διαδικασία ε, γιατί στις διαδικασίες επιλογής δηλαδή στις επιτροπές ε, ορισμένοι διακυβεύουν και την ίδια τους την υπόσταση και τη φήμη όταν συμμετέχουν σε τέτοιες διαδικασίες ε, και δεν θέλουν πια να συμμετέχουν. 44 είναι ε, στη Γενική Διεύθυνση 22, 25 και 29 στις διευθύνσεις. Αυτό το εννοείται, είστε σοβαροί, θα παραμείνει έτσι ή θα το αλλάξετε. Ε, ε, θα κόψετε με συγχωνεύσεις καμιά υψηλή θέση για να υπάρχει και μία αντιστοιχία των θέσεων αυτών μεταξύ των διαφόρων θεσμικών οργανών προς το οργανόγραμμα. Ε, μιλώ για τις υψηλέ θέσεις. Το επόμενο θέμα. Για μένα θα είχε σημασία να προωθηθεί αυτή η πρωτοβουλία για τις έξυπνες οικονομίες. Αυτό το smart savings το έχετε ποσοτικοποιήσει, το έχετε υπολογίσει. Καλό είναι και μ' αρέσει και θέλω να το υποστηρίξω. Είναι πάρα πολύ ωραία πρωτοβουλία και αξιολογή. Αλλά το έχετε μετρήσει τι θα βγει από αυτό. Και επίσης κάτι άλλο σημαντικό. Να μας δώσετε την κατανομή των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου. Εσείς δεν κάνετε μόνο διοίκηση, έχετε και πολιτικές αρμοδιότητες. Οι άλλοι τι κάνουν οι υπόλοιποι εκτός από εσά. Λαμβάνουμε υπόψη μας τις απαντήσεις που μας δίδονται, αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να έχουμε σε ένα χαρτί το οργανόγραμμα, την κατανομή αρμοδιοτήτων, ποιος είναι αρμόδιος γιατί, για να ξέρουμε πού πηγαίνουμε. Μετά, έχουμε μια πολύ περίεργη, μια μυστήρια υπόθεση. Στις εκθέσεις των πρέσβεων είδαμε το, το 57% να λέει ότι θεωρούν τους συνεργάτες τους περιορισμένων προσόντων. Όλοι ακολούθησαν κάποια προγράμματα κατάρτισης εκπαίδευσης, 57% των πρέσβεων λένε ότι δεν οδήγησε πουθενά. Γιατί το κάνουμε. Μπορείτε να μας δώσετε στοιχεία γι' αυτό. Αυτό φορά και η δερμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι και προσωπικό της ΔΕΒΚΟ αλλά όταν τόσοι πολλοί πρέσβες δηλώνουν τέτοια πράγματα δεν μπορεί να μας είναι αδιάφορο ούτε εσάς. Ε, θα παρακαλούσα επίσης το ελεκτικό συνέδριο να μας απαντά στις ερωτήσεις μας και στην ειδική του έκθεση περισσότερο να μας πει ποιο είναι το κόστος πρόσληψης. Δηλαδή, Πόσο κοστίζει να προσλάβει κάποιο ε, ή να αποσπάσει ένα πρέσβη κράτου μέλου. Τι κοστίζει να αποσπαστούν οι πάλι τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή με συγκεκριμένα στοιχεία. Επίσης, στην ειδική έκθεση το ελεκτικό συνέδριο να ασχοληθεί και με το οργανόγραμμα στα κεντρικά γραφεία, στην έδρα της ΙΕΒ. Πώς είναι οργανωμένο. Υπάρχουν αρμοδιότητες διπλές επικαλύψεις. Γιατί ακούμε από την οργάνωση. Και εσείς είστε πολύ παλιά καραβάνα κύριο Σάλιβαν και τα γνωρίζετε αυτά πάρα πολύ καλά. Επίσης το ελεκτικό συνέδριο να κοιτάξει και τους ειδικού εντεταλμένους και τους ειδικού απεσταλμένους και το κόστος ε, και να το συγκρίνει με τη σημασία και τη σκοπιμότητα της θέσης. Ευχαριστώ κύριο Βόν. <clears throat> Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε θεωρώ ότι όσον αφορά την υπηρεσία, πρόκειται για μια νέα υπηρεσία και κάνει εξαιρετικό έργο τόσο το, έργο, το ίδιο το έργο όσο και ο χειρισμός του προπολογισμού κατά το πρώτο έτος λειτουργίας. Σε αυτό το πρώτο έτος ε, σίγουρα είχατε να αντιμετωπίσετε πολλές προκλήσεις όσον αφορά το προσωπικό, τη σωστή εξισορρόπησή του, ότι πήρατε ένα απερχαιωμένο σύστημα πληροφορικής από το Συμβούλιο, ότι έπρεπε να διασφαλίσετε ασφαλή κτίρια σε κάποια επικίνδυνα μέρη του κόσμου, μεγάλες προκλήσεις δηλαδή. Θα θέλαμε να μας πείτε λοιπόν πώς αντιμετωπίσατε αυτές τις προκλήσεις και κατά πόσο έχετε την αίσθηση ότι έχετε λύσει όλα τα προβλήματα. Και το τελευταίο που θέλω να πω σχετίζεται με κάτι που παρατηρήσα όταν ασχολήθηκα με τον προπολογισμό άλλων τμήματων για το 2013. Ξέρετε ότι ήμουν εισηγητή για κάποια άλλα τμήματα και κάτι που με έκανε εντύπωση είναι η έκθεση που πόσο είστε εκτεθειμένοι σε ορισμένες ε, αυτομοιώσεις ε, κατά πόσο αισθάνεστε ότι στο μέλλον θα μπορούσατε να μειώσετε αυτή την έκθεση. Ευχαριστώ, Παλ Ρούμπιχ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι εμείς εδώ στην Ευρώπη ε, κάναμε ένα σημαντικό βήμα και στις διεθνείς σχέσεις μας αντίστοιχα έχουμε δυνατότητες διαμόρφωσης αυτών. Ένα από τα βασικά προβλήματα στην Ευρώπη αυτό τον καιρό είναι η ενεργεία και ιδιαίτερα η ενεργεία των νέων. Θα μπορούσατε να φανταστείτε η υπηρεσία εξωτερικής δράσης να ειδικευθεί κάπως περισσότερο να εξειδικευθεί στις οικονομικές εξωτερικές μας σχέσεις, ιδιαίτερα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Να έχουν ένα συνομιλητή εκεί ε, για να ε, μπορούν να ενημερώνονται, να έχουν επαφές και κυρίως οι ευρωπαϊκές πρεσβείες να αναλάβουν ένα ρόλο συντονιστικό μεταξύ των κρατών μελών για να αυξηθεί το δυναμικό εδώ που προσφέρεται στην Ευρώπη και να υπάρχουν ενδεχομένω και ανταλλαγέ νέων, έτσι με τρόπο πιο εντατικό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σόνικ τελευταίος αυτό το γύρο. Mm, Ευχαριστώ πολύ η κυρία Άστον παρουσίασε τον κύριο Σάλιβεν ως εμπειρογνώμονα σε θέματα για τη Ρωσία επίσης. Ήθελα λοιπόν να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία για να κάνω μερικές ερωτήσεις. η ΑΕΔ υποστηρίζει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη διένεξη μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Gazprom στη Ρωσία όσον αφορά το, πακέτο, το ενεργειακό πακέτο και άλλες δραστηριότητες σε αυτόν τον τομέα. Ποιες είναι οι απόψεις σας, πώς προβλέπετε το μέλλον όσον αφορά αυτή τη διαφορά. Και δεύτερον, ε, ένας Πολωνός, ε, ο Πολωνός Υπουργός Εξωτερικών επικοινώνησε πρόσφατα με την κυρία Άστον ζητώντας βοήθεια για την περισυλλογή των συντριμιών του αεροπλάνου του Πόλεφ όπου σκοτώθηκε ο πρόεδρος της ε, Πολωνίας κατά τη συντριβή του και η Ρωσία δεν θέλει να δώσει αυτό το αυτά τα συντρίμια στη προηγούμενη σύνοδο κορυφής μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας αναφέρθηκε αυτό το ζήτημα. Η υπηρεσία σας θα εξακολουθήσει, θα συνεχίσει τις πιέσεις ώστε να καταλήξουμε σε θετικό αποτέλεσμα. Γι' αυτό το έθιμα ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ τους συναδέλφους όλους για τις ερωτήσεις τους και θα παρακαλούσα τώρα τον κύριο Σάλιβαν να απαντήσει. Είναι ο διοικητικός γενικός διευθυντής της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στα διάφορα σημεία που αναφέρθηκαν. Αναγνωρίζω φυσικά ότι δεν μπορώ να αντικαταστήσω επαρκώς την ε, είπατε εκπρόσωπο. Κύριε Οντή, όσον αφορά την ερώτησή σας ε, για την περίμετρο της συζήτησης, το πεδίο της συζήτησης, η ερώτησή σας είναι περισσότερο πολιτική και όχι γραφειοκρατική. Η γραφειοκρατική απάντηση είναι ότι εδώ είμαστε για να δώσουμε λογαριασμό για τη διαχείριση του ε, διοικητικού προϋπολογισμού της ΕΕΔ και τα κονδύλια που διαχειρίζεται η υπηρεσία εξωτερικής πολιτικής. Αυτά είναι τα κονδύλια για τα οποία επίσημα είμαστε υπεύθυνοι. Μα ζητείτε να δώσουμε απαλλαγή για το διοικητικό προπολογισμό. Έχουμε... Η, η, η δεν είναι νέος θεσμός. Πάντα το λέω Είμαστε ναι, υπηρεσία για δύο λόγους, για να μπορείτε να μας ελέγχετε σε δημοσιονομικά θέματα, να είμαστε υπόλογοι προς εσάς ως προς τη δαπάνη των κονδυλίων και η κυρία Άστον έχει αυτονομία όσον αφορά τη διαχείριση του προσωπικού. Κατά τα άλλα δεν είμαστε ε, θεσμικό όργανο, πρέπει να συνεργαζόμαστε στενά με τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα. Η συζήτηση λοιπόν αφορά το διοικητικό μας προπολογισμό. Και ευχαριστώ το ελεκτικό συνέδριο για τα όσα είπε και αναμένουμε τα αποτελέσματα ε, της αξιολόγησης τους ε, όσον αφορά την επίδοση των δομών μας. Χαίρομαι που τουλάχιστον για φέτος δεν βρήκαν ε, υλικά λάθη στη δημοσιονομική μας διαχείριση μέχρι στιγμής. Εδώ και καιρό ασχολούμαι με αυτά τα ζητήματα και γνωρίζω ότι στη δημοσιονομική διαχείριση είσαι τόσο καλός όσο η τελευταία αξιολόγηση και η διαδικασία διατήρησης των, του επίπεδου που θέλουμε είναι συνεχής. Πιστεύω ότι μπορούμε να σας διασφαλίσουμε επαρκώς για, τα, για τις δομές μας, αλλά μερικές φορές σε επικίνδυνα περιβάλλοντα, σε μακρινά ε, χώρες δεν είναι εύκολο να έχουμε πλήρη έλεγχο. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να συνεχίσουμε να επιδιώκουμε, να διατηρούμε τα υψηλά πρότυπα Όσον αφορά την πρόταση σας για οικονομικό έλεγχο, κύριε Όντι, θα το κρίνετε εσείς ε, και το ελεγκτικό συνέδριο, αλλά εγώ θέλω να είμαι σαφής. Ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα της δημιουργίας αυτής της υπηρεσίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τα κράτη-μέλη είναι ότι αλλάζει το περιβάλλον των διμερών δραστηριοτήτων των κρατών μελών. Δεν αντικαθιστούμε τα κράτη-μέλη. Παρέχουμε δυνατότητα μεγαλύτερων συνεργειών. Πιστεύω έχετε δίκιο. Η συνεργασία μας σε τρίτες χώρες, η συστέγαση σε ιδιακτήρια, η, η χρήση ίδιων διοικητικών δαπανών, αυτό είναι το μέλλον και πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι που το επιθυμούν τα κράτη-μέλη. Είναι εύκολο στα λόγια, αλλά πολύ πιο δύσκολο στις πράξεις. Εγώ έχω δεσμευτεί γι' αυτό, αλλά θα σας διαβεβαιώ, μιλώντας με συναδέλφους έμπειρους στα κράτη-μέλη, για παράδειγμα από τις σκανδιναβικές χώρες, ε, Τι χώρες του Μπενελούξ Επίση, ε, αυτό έχει γίνει εκτενού. θα σα πούν όλοι αυτοί ότι η δραστηριότητα αυτή είναι επικίνδυνη θέλει συγχρονισμό κτίριων δραστηριοτήτων ε, ορών λειτουργία, επίπεδα στελέχωση και ούτω αλλά έχουμε δεσμευτεί απόλυτα σε κάθε πρωτεύουσα όπου έχουμε παρουσία να συνεργαζόμαστε στενά με τα κράτη-μέλη, να δίνουμε ευκαιρίε για συνέργειε όπω κάναμε με την Ισπανία, όπω αναφέρθηκε, όταν μείωσε τον αριθμό στελεχών τη, των αποστολών τη η Ισπανία ε, χρησιμοποίησαμε Ισπανούς διπλωμάτες ε, να λειτουργήσουν στο πλαίσιο των αντιπροσωπιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο Χοτσιμίνγκ, στο Βιετνάμ θέλουμε να συγκεντρώσουμε τις προξενικές υπηρεσίες των κρατών μελών ώστε να υπάρχει ε, ένα ενίο σημείο εξυπηρέτηση για την παροχή θεωρήσεων για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες και ελπίζω ότι, και πιστεύω ότι σε 4-5 χρόνια δεν θα όχι σε 12 μήνε βέβαια, θα μπορούμε να επανέλθουμε σε αυτό το κοινοβούλιο και να έχουμε αποδείξει ότι έχουμε αλλάξει τον τρόπο διεξαγωγής δραστηριοτήτων μεταξύ των αντιπροσωπιών των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς όφελος τόσο του φορολογουμένου, του Ευρωπαίου και του Εθνικού Φορολογουμένου. Θα ήθελα λοιπόν πολύ να προχωρήσουμε τις εργασίες μας και να δούμε πώς θα μπορούσαμε να επιτύχουμε καλύτερα αποτελέσματα πιο γρήγορα. Έχουμε δεσμευτεί ενεργά ε, με τα κράτη-μέλη. Ο Βανσό, που είναι διευθυντή προπολογισμού, έχει συμμετέχει σε πολλέ συνεδριάσει με πολύ κόσμο από τι εθνικέ υπηρεσίε σε θέματα διαχείριση κτηρίων και σχεδιασμού της μελλοντική επέκταση του δικτύου. Όσον αφορά την πολυγλωσία, το σημειώνω Νομίζω διαφορετικά για την ιστοσελίδα, αλλά το λαμβάνω πολύ σοβαρά. Έχετε δίκιο και ξέρετε ότι αντιμετωπίζω πολύ σοβαρά το ζήτημα τη πολυγλωσία στην Ευρώπη. Αποτελεί ένα από τα ισχυρά σημεία τη Ευρωπαϊκή Δημοσίας και πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για αυτό. Όσον αφορά την κινητικότητα, κύριε Μαγιάλα, ε, είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα. Τι κάνουμε στην ΕΕ, συγχρονίζουμε, έχουμε μια ενοποιημένη διαδικασία κινητικότητας. Κάθε χρόνο το 1 τέταρτο του προσωπικού μας στις αντιπροσωπείες μετακινείται, διότι αποσπώνται για τέσσερα χρόνια το προσωπικό. Κάθε τέσσερα χρόνια λοιπόν το 1 τέταρτο μετακινείται. Τι κάναμε εμείς Υιοθετήσαμε παρόμοια διαδικασία κινητικότητα στα κεντρικά. Λέμε ότι όταν κάποιο εργάζεται για τέσσερα χρόνια σε μία θέση στα κεντρικά, τότε μετακινείται. Συγχρονίζουμε δηλαδή τη μετακίνηση στα κεντρικά μα και στι αντιπροσωπείε μα. Αυτό δημιουργεί πολύ μεγαλύτερε δυνατότητε για όσου επανέρχονται από, από τι αντιπροσωπείε να βρουν μία θέση στα κεντρικά και ενθαρρύνουμε του όσου εργάζονται στα κεντρικά να καταλάβουν ότι αν θέλουν σταδιοδρομία σε μια διπλωματική υπηρεσία θα πρέπει να υπηρετήσουν και σε μια αντιπροσωπεία. Δεν ήταν απαραίτητα αυτή η φιλοσοφία της Γενικής Διεύθυνσης Εξωτερικών Σχέσεων, αλλά αυτή είναι η κατεύθυνση, πιστεύω, προς την οποία πρέπει να κινηθούμε. Αυτό που φυσικά πρέπει να εξορροπηθεί και με την απόκτηση δεξιοτήτων, γνώσεων. Πρέπει να είμαστε κάπως ευέλικτοι. Δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε κάτι τέτοιο με απόλυτη αυστηρότητα, διότι δεν θέλουμε να χάσουμε ε, εκπροσώπους σε κρίσιμες στιγμές διαπραγμάτευσης, αλλά θεωρητικά κάθε τέσσερα χρόνια οι άνθρωποι αλλάζουν δουλειά και μετακινούνται μεταξύ κεντρικών γραφείων και αντιπροσωπιών. Κύριε Σαλαφράνκα, όσον αφορά τις ε, εκλογικές αποστολές, έχει γίνει εκτενής αξιολόγηση του κόστους κάθε εκλογικής αποστολής με το λεπτομερές δημοσιονομικό εργαλείο και φυσικά μπορούμε να το συζητήσουμε μαζί σας, είμαστε στη διάθεσή σας. Ένα από τα μεγάλα κόστη είναι συνήθως η ασφάλεια διότι πολύ συχνά οι αποστολές αυτές ε, λαμβάνουν χώρα σε δύσκολο ε, πολιτικό περιβάλλον. Σίγουρα θα σας δώσουμε περισσότερες πληροφορίες εφόσον το επιθυμείτε όσον αφορά το ποσοστό του ανώτερου προσωπικού όπως αναφέρθηκε από την κυρία Γκρέσλε. Κοιτάξτε, το σημειώνω. Πιστεύω ότι οι πρακτικές μας δεν διαφέρουν υπερβολικά από τις πρακτικές των κρατών μελών. υπάρχουν συχνά ανώτερα στελέχη. Πρέπει να βλέπουμε την ισοτιμίωση και τη δυνατότητα ε, ε, συνεννόησης των ανθρώπων αυτών με διπλωμάτες ξένων χωρών σε αυτόν τον κόσμο της διπλωματίας. Και οι βαθμοί και οι τίτλοι ε, κάνουν μια διαφορά. Φυσικά έχουμε κληρονομήσει μια κατάσταση όπου έχουμε σχετικά γυρεότερους αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έρχονται από τη Γραμματεία του Συμβουλίου είτε από την Κομισιόν και αυτοί οι άνθρωποι έχουν τους βαθμούς που έχουν. Το κληρονομίζαμε αυτό το προσωπικό ε, κοιτώντας τη δημογραφική κατάσταση της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Υπηρεσίας ε, κάθε χρόνο βλέπουμε όλο και περισσότερο να παίρνουν σύνταξη και μετά να έρχονται νεότεροι άνθρωποι αλλά είναι ένα σημείο το, στο οποίο είμαστε ευαισθητοί και το εξετάζουμε τώρα. Όσον αφορά το κόστος και το ωφέλη, με συναδέλφου τη ΔΕΒΚΟ κάναμε μια αξιολόγηση όπου εξετάσαμε λεπτομερώ τη στελέχωση της Κομισιόν και της ΔΕΒΚΟ στι δικές μας αντιπροσωπείες ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι αξιοποιούμε σωστά τα χρήματα. Διότι στην Ασία και στη Λατινική Αμερική. Ας πούμε σήμερα ξοδεύουμε λιγότερα χρήματα στην Αφρική, για παράδειγμα περισσότερα όσον αφορά την αναπτυξιακή πολιτική που εστιάζεται στις φτωχότερες χώρες. Η ΔΕΦΚΟ αυτή τη στιγμή προσαρμόζει την παρουσία της στις αντιπροσωπείες ώστε να προσαρμοστεί. Και εμείς διεξάγουμε αυτό που λέμε zero-based review ώστε να δούμε κατά πόσο υπάρχει περιθώριο, κατά πόσο έχουμε τους σωστούς ανθρώπους στις σωστές θέσεις Δυστυχώς το συμπέρασμα είναι ότι έχουμε ανεπαρκή στελέχωση, τουλάχιστον σε επίπεδο πολιτικού προσωπικού και ατόμων που έχουν αναλάβει τα νέα καθήκοντα που έχουμε αναλάβει ως Ε.Ε.Δ. δεν έχουμε αρκετό κόσμο για να κάνει όλα τα πράγματα που θα θέλαμε. Μελετάμε για να δούμε πώς θα λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Κυρία Γκρέσλε, όσον αφορά το ζήτημα του κόστους πρόσληψης, δεν μπορώ να σας δώσω αυτή τη στιγμή ένα αριθμό, αλλά να το εξετάσουμε. Φαντάζομαι μπορούμε να, να δούμε πόσο κοστίζει η διαδικασία προσλήψεων. Πρέπει να καταλάβετε ότι η περίοδος που περάσαμε μόλις τώρα ήταν εξαιρετική κατά κάποιο τρόπο. Δεν πρόκειται να επαναληφθεί σύντομα. Χρειάστηκε να δημοσιεύσουμε πάρα πολλές θέσεις, ε, είχαμε πάρα πολλούς υποψήφιους. Ήταν κάπως ε, εξαιρετική αυτή η περίπτωση. Αφού μπούμε σε μια τροχιά, δεν θα χρειάζεται να εφαρμόζουμε τόσο εντατικέ ε, διαδικασίε ε, πρόσληψη. Τώρα, όσον αφορά την αποτελεσματικότητα και τη διαφάνεια τη διαδικασία προσλήψεων, θα το κρίνουν άλλοι και μπορούν να επικρίνουν άλλοι. Αλλά εγώ το μόνο που μπορώ να σα πω είναι ότι συνεργαστήκαμε στενά με τα κράτη-μέλη και με την Επιτροπή και με την Γραμματεία του Συμβουλίου σε ομάδε εργασία, στι διαδικασίε, στην διεκπαιρέωση, στη των αιτήσεων, στις συνεντεύξεις και ειλικρινά είχα ζητήσει σχόλια από όλους και όλοι είπαν εργαζόμαστε επαγγελματικά και αντικειμενικά όσον αφορά αυτή την πολύπλοκη διαδικασία προσλήψεων. Άλλες προτάσεις, άλλες κάποιες, κάποιοι που λένε ότι κάποιοι είχαν, ε, ήταν φωτογραφικές οι θέσεις τους ε, ορισμένοι απλά ήταν υπερβολικά καλοί υποψήφοι και φανταζόμασταν από την αρχή ποιον θα προσλαμβάναμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα περάσουμε τη διαδικασία, δεν θα εφαρμόσουμε μια διαφανή διαδικασία επιλογής. Πιστεύω λοιπόν ότι γενικά έχουμε κάνει έργο με διαφάνεια, αλλά φυσικά πάντα θα επικρίνεται Είναι προτιμότερο λοιπόν να ε, εφαρμόσουμε και να δώσουμε και χρήματα για αυτές τις εξοικονομήσεις. Χρειάζονται αλλαγές σε κάποιους κανονισμούς. Στον ιστορικό κανονισμό προσωπικού εξετάζουμε σοβαρά το ζήτημα του δικαιώματος αναχώρησης, τις κατοικίε. Προσπαθούμε να εφαρμόζουμε τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα προς το κόστος και προσπαθούμε να βρούμε τρόπους να εξοικονομήσουμε χρήματα, να είμαστε πιο αποτελεσματικοί ως προς το κόστος και θα σας αναφέρουμε τα αποτελέσματα του όλου εγχειρήματο. Όσον αφορά την κατανομή αρμοδιοτήτων, εσωτερικά έχουμε έγγραφα που το εξηγούν. Ευχαρίστω για λόγους διαφάνειας θα, σας θα, θα τα θέσω στη διάθεσή σας. Φυσικά κανένα γραφειοκρατικό σύστημα δεν μπορεί να περιγράψει ακριβώς πώς λειτουργούν τα πράγματα στην πραγματικότητα, αλλά ε, εμείς γνωρίζουμε ποιο κάνει τι. Τώρα όσον αφορά την επίκριση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τα νούμερα έχουν συγκεντρωθεί από του συναδέλφου μας στην ΤΕΒΚΟ και πιστεύω ότι η κατάρτιση όντω είναι πολύ σημαντικό ζήτημα και πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να, είναι, να λειτουργεί ορθά. Κύριε Βόν, όσον αφορά τις προκλήσεις, ε, ευχαριστώ πολύ που μου κάνετε την ερώτηση. Η μεγαλύτερη πρόκληση ήταν ότι έπρεπε να συστήσουμε τα δικά μας συστήματα δημοσιονομικού, δημοσιονομικής διαχείρισης, διαχείρισης προσωπικού, οικονομικού ελέγχου, προστασίας δεδομένων, πρόσβαση στα έγγραφα, όλα τα εργαλεία του ενός οργάνου, ενός θεσμικού οργάνου. Έπρεπε να τα δημιουργήσουμε μόνοι μας κατά τη σύσταση της υπηρεσίας. Δεν ήταν κάτι εύκολο δεδομένου ότι είχαν ξεκινήσει οι δραστηριότητες μας και ότι ταυτόχρονα έπρεπε να τα σε κρίσει και να εφαρμόζουμε πολιτικές. Τώρα όσον αφορά τι διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, όταν πέφτει το ευρώ κατά 5% σε σχέση με το δολάριο, αυτό μας ε, κοστίζει 250 εκατομμύρια ευρώ. Τόσο πολύ επηρεάζουν οι διακυμάνσεις ε, ε, των συναλλαγματικών ισοτιμιών το έργο μια υπηρεσία σαν τη δική μα. Δεν είμαστε οι μόνοι και οι διπλωματικέ υπηρεσίε αντιμετωπίζουν την ίδια πρόκληση. Ότι χρειάζεται κάποια ευελιξία δημοσιονομική ώστε να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα των συναλλαγματικών ισοτιμιών που επηρεάζουν τα κόστη μα. Κύριε Ρούμπικ, όσον αφορά τη μεγαλύτερη πρόκληση είναι η οικονομική. Έχετε απόλυτα ζήτημα. Η ανεργία των νέων είναι ένα από τα σοβαρότερα ζητήματα με σημαντικές κοινωνικές επιπτώσεις. Εγώ πιστεύω ακραδάντα ότι χρειαζόμαστε περισσότερη ευρωπαϊκή δέσμευση στην παγκόσμια οικονομία. Το μεγαλύτερο κομμάτι της ανάπτυξης για την Ευρώπη θα έρθει εκτός Ευρώπης και πρέπει να υποφεληθούμε, να το αξιοποιήσουμε με την εμπορική μας πολιτική οι αντιπροσωπείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεργάζονται στενά με τις επιχειρήσεις ε, στις διάφορες χώρες ε, όπως έχουμε τα επιμελητήρια στο Πεκίνο, στο Τόκιο, στο Βιετνάμ όπου δημιουργείται αυτή τη στιγμή συνεργαζόμαστε στενά με ευρωπαϊκά επιμελητήρια τοπικά ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι μιλάμε ε, ε, εξ ονόματι των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και ότι τις βοηθάμε, αλλά να βοηθήσουμε και τις εταιρείε που θέλουν να μπουν σε αυτές τις αγορές και η Γενική Διευθύνση Εμπορίου έχει ένα πολύ καλό σύστημα πρόσβασης στις αγορές που ενημερώνει ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ε, οι οποίες προσπαθούν να δραστηριοποιηθούν σε ξένες αγορές. Εμείς έχουμε δεσμευτεί και εγώ έρχομαι σε επαφή με το Business Europe, με διάφορα επιμελητήρια ώστε να φροντίσουμε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική δράση να βοηθάει τι ευρωπαϊκέ επιχειρήσει και το ευρωπαϊκό εμπόριο ώστε να υποφεληθούν από τι εμπορικέ ευκαιρίε που υπάρχουν εκεί και Ο πρόεδρος του Business Europe ζητήθηκε από την κυρία Καθρινάστον να μιλήσει το Σεπτέμβριο στο συνέδριο που είχαμε. Μίλησε εκεί, εκτιμήθηκε ιδιαίτερα η παρουσία του και η δυνατότητα που είχε να ε, μιλήσει με του πρέσβει μα Όσον αφορά τη Ρωσία κύριε Πρόεδρε, θα απαντούσα τώρα την ερώτησή σας για τη Ρωσία. Ενημέρωσα την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων χθε στη Σύνοδο Κορυφή. Το ζήτημα τη ενέργεια ε, είναι ιδιαίτερα επίμαχο σχέση μα με τη Ρωσία. Το τρίτο ενεργειακό πακέτο, όπω ξέρετε, αμφισβητείται από του Ρώσου συναδέλφου. Εμεί ακολουθήσαμε σκληρή γραμμή στη Σύνοδο Κορυφή ότι θα εφαρμοστεί το τρίτο ενεργειακό πακέτο σε όλη την επικράτεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση. η ευελιξία αυτού του πακέτου θα μπορέσει να βοηθήσει σε εξαιρετικέ περιπτώσει, βέβαια, αλλά εμεί δώσαμε ένα σαφέ μήνυμα ότι η Gazprom και οι άλλοι Ρώσοι φορεί θα πρέπει να συμμορφωθούν με του κανόνε ενιαία αγορά. Δεν συζητήσαμε την περίπτωση antitrust, διότι αυτό είναι θέμα επιχειρησιακής, ε, επιχειρησιακού απορρίτου. Αυτό πρέπει να το χειριστεί η Γενική Διευθύνση Ανταγωνισμού, όπως κάνουμε και έρευνες ε, κατά άλλων εταιριών, όπως για παράδειγμα η Microsoft. Ε, γνωστό παράδειγμα. Δεν μπορούν λοιπόν να μας κατηγορήσουν οι συνάδελφοι ότι θυματοποιούμε μια εταιρεία και όχι μια άλλη. Όσον αφορά για τη Σαρία, προσπαθούμε πάντα να παρέμβουμε ώστε να υποστηρίξουμε τα κράτη-μέλη μας που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα προβλήματα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, αλλά σε ορισμένα Εάν μα ζητάει ένα κρατός μέλος να βοηθήσουμε σε κάποιο εθνικό πρόβλημα μια τρίτη χώρα, προσπαθούμε πάντα να παρέχουμε τη μέγιστη υποστήριξη και αρρωγή. Και αυτό έκανε και η καθήση σε αυτή την περίπτωση. Θα συνεχίσουμε λοιπόν να παρέχουμε αυτή την υποστήριξη όταν χρειάζεται. Κύριε Πρόεδρε, ελπίζω να κάλυψα τα περισσότερα ζητήματα. Είναι πολλά τα ζητήματα. Με μεγάλη ευχαριστή θα συνεχίσουμε αυτόν τον πολύ καλό πιστεύω διάλογο με τα μέλη, με τον κύριο Σιγητή, ώστε να μπορέσουμε να συμπληρώσουμε τι πληροφορίε, όπω εσεί θα κρίνετε απαραίτητο σε γραπτή ή άλλες μορφές μετά από τη σημερινή συνάντηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε να δείτε. Έχουμε δύο συναδέλφους οι οποίοι έχουν ζητήσει το λόγο. Έχει το λόγο. Η κυρία Κρέσλερ και μετά ο κύριος ε, Πίνξτεν. Κύριε Πίνξτεν, θέλετε να απαντήσετε. Ναι, ευχαριστώ πρόεδρε. Να απαντήσω εν συντομία σε δύο κοινά. Για το δεύτερο θέμα, ε, δώσατε τον λόγο, εάν θελήσετε, στον κύριο Τομέ, τον συναδελφό μου. Το πρώτο που θέλω να ρωτήσω είναι το εξή. Όταν ελήφθη η απόφαση στο Ελληνικό Συνέδριο να κάνουμε αυτόν τον έλεγχο όσον αφορά την υπηρεσία, ε, συζητήσαμε στα δύο τμήματα. Πρώτα πρώτα στο υπαριθμό 3, το υπεύθυνο που αυτό που ασχολείται με την εξωτερική πολιτική και επίση και στο τμήμα του Ελληνικού Συνεδρίου όπου εργάζεται ο κύριο Τομέ. Το υπαρθμόν 4. Ε, αυτό το τμήμα του Ελληνικού Συνεδρίου ασχολείται με παντό είδου δαπάνη. Τελικά όμω συμφωνήθηκε από τα δύο τμήματα να γίνει ένα και μόνο έλεγχο. Οπότε με αυτόν τον έλεγχο θα καλύψουμε όλα όσα αφορούν τις διοικητικές δαπάνες και είπαμε για αυτόν τον λόγο να έχουμε κάποιο είδους ε, σφαιρικό, γενικό έλεγχο ε, μέχρι σήμερα δεν αποφασίσαμε πάντως στο τρίτο τμήμα ακριβώς τι εύρος, τι βεληνικές θα έχει αυτός ο έλεγχος. Ε, αλλά βέβαια είπαμε ότι θα καλύψουμε και θέματα πολιτικής αλλά και τις ε, δαπάνε. δαπάνες. και τα μεν και τα δε θα τα καλύψουμε τον εχθρό. Αυτά έχω να απαντήσω στην κυρία Γκρέσλα. Ποιος μου γρούθα τώρα. Εάν ε, συμφωνείτε κύριε Πρόεδρε θα μπορούσε να διεξέλθει τα επόμενα από όσα ήθελε να διευκρινίσει η κυρία Γκρέσλε. Ε, ε, Μου ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτα πρώτα θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ακριβώς ποιο θα είναι το βιλινικές του έργου το οποίο θα επιτελέσουμε ή επιτελούμε ήδη στο ελεγκτικό συνέδριο για τις διοικητικές δαπάνες. Κοιτάξτε, έχουμε το κεφάλαιο υπαριθμών 9 στην έκθεση αυτή. Εκεί εξετάζουμε τα των διοικητικών δαπανών για όλες τις υπηρεσίες, όλα τα θεσμικά όργανα. Και η ΑΕΡ είναι ένα από αυτά τα και είπαμε επομένω το 2012 οι δαπάνε ε, και, και οι σχετικέ καυρίτσε δεν έπασχαν κάποιο τυπικό σφάλμα. Είπαμε ε, ο ρυθμό, τέλο πάντων το, το, το, των σφαλμάτων γενικά ε, για την ΕΕΔ ανέρχονταν στο 0,1%. από τι 5 αλλαγές βρήκαμε 4 λάθη και αυτό ήταν λοιπόν το 0,1%. Επίση ασχοληθήκαμε και με έλεγχο των συστημάτων Βρήκαμε όμω και κάποια σημεία τα οποία έπασχαν για την ΕΕΔ, ακριβώς όπως το τόνισε ο Γιώργος Πίνξτεν, ο συνάδελφος, Οπότε και διατυπώσαμε τις σχετικές συστάσεις επιπλέον. Είχαμε αυτές τις ε, ειδικέ συνθήκες ε, που συντρέχουν και λήφθησαν υπόψη σε σχέση με την υγεία Και έτσι θα συνεχιστεί η ανάλυση μας επί τη βάση των προηγουμένων οικονομικών ελέγχων των ιστορικών ελέγχων και των εκθέσεων δραστηριοτήτων από τις διάφορες υπηρεσίες. Πάλι σχετικά με την ΑΕΔ, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει κάποιο κίνδυνο σε σχέση με τις ειδικέ συνθήκες τη λειτουργία. της ΑΕΔ. Όπως είπαμε προηγουμένως, παρά τόσο έχουμε συμφωνηθεί από τις γενικές διευθύνσεις, διάφορες υπηρεσίες, γιατί είναι αρκετά δύσκολο κανείς να κάνει αυτό που κάνει η ΕΕ. Οπότε, και ακριβώς λάβουμε υπόψη τις δυσκολίες που έχουν δημιουργήσουν οι αντιπροσωπείες που δρούν σε ξένο περιβάλλον. Ευχαριστώ. Έχουμε άλλους τρεις που θα κάνουν ερωτήσεις στον κύριο Σάλιβαν, ο κύριος Σικέρσκι, ο Κύριο Οντί και η κυρία Γκρέσλε. Ε, Για να ολοκληρωθεί η συζήτηση. Ο κύριος Σικέρσκι πρώτος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μια σύντομη ερώτηση έχω εγώ. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, ε, μεταξύ των εργαζομένων σας, έχετε εκπροσώπους από ε, μια συγκεκριμένη θεματική ε, υπηρεσία. Δηλαδή, εκείνος που ασχολείται με την ενέργεια στη συνεργασία με τη Ρωσία είναι αποσπασμένος υπάλληλο ή διορισμένος ε, από το αντίστοιχο θεματικό πλαίσιο, από την αντίστοιχη υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ασχολείται αποκλειστικά με την ενέργεια. Υπάρχει αυτή η σχέση με το περιεχόμενο οι εμπειρογνώμονες απασχολούνται ε, για τα θέματα τα οποία είναι ειδικοί. Γιατί το ρωτάω. Γιατί ξέρω ότι υπάρχουν στι υπηρεσίε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή άριστοι και πάρα πολύ καταρτισμένοι υπάλληλοι που ασχολούνται με αυτά τα θέματα. Για τη συγκεκριμένη περίπτωση της Ρωσίας, ε, ο αρμόδιος ε, για αυτά τα θέματα είναι ο ειδικό. Καλό θα ήταν λοιπόν να μας απαντήσετε σε αυτό. Ο κύριος Σοντή, ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, ε, συγγνώμη που επιμένω, αλλά ακόμα δεν κατάλαβα ποια είναι η περίμετρο του λογιστικού ελέγχου. Θα ήθελα να μάθω τι ελέγχουμε εμείς στο Κοινοβούλιο, εμείς οι βουλευτές. Ε, ο στόχος του Κοινοβουλίου σε κάθε δημοκρατία είναι να ελέγχει την εκτελεστική εξουσία και να υπάρχουν και κυρώσεις. Ε, παράδειγμα, αν αρνηθούμε την απαλλαγή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε δυσπιστία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να την απολύσουμε εμπολή. Εγώ ακόμα δεν κατάλαβα τι ελέγχουμε εδώ. Ο κύριος ο Σάλιβαν μας είπε, αν κατάλαβα καλά, ότι η απαλλαγή μας αφορά τις ε, διοικητικές δαπάνες, τις λειτουργικές. Μάλιστα. Ε, τρία είναι τα μέλη του ελεκτικού συνεδρίου που έχουν άποψη για τις λειτουργικές αυτές, αλλά και για τις επιχειρησιακές δαπάνες ε, ένας λογιστικός έλεγχος για τρεις επιτρόπους και για διοικητικές και για επιχειρησιακές δαπάνες. Αυτό πώ γίνεται. εμεί τι ψηφίζουμε από όλα αυτά, τι θα συστήσουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σα συνιστούμε την απαλλαγή επιπίου αντικειμένου. Αυτό δεν το έχω καταλάβει. Ε, γιατί ε, θα ακολουθήσουν και άλλες απαλλαγές στο μέλλον και η επόμενη διαδικασία θα είναι η τελευταία πριν τις ευρωπαϊκές εκλογές και επειδή οι πολίτες μας ρωτούν τι κάνατε από πλευράς δημοσιονομικού ελέγχου. Εμείς τι θα ψηφίσουμε, για ποιες δαπάνες δίνουμε απαλλαγή ή όχι. Ευχαριστώ κύριε Γκρέσλε για την τελευταία ερώτηση. Λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά θα πρέπει να ξεκαθαρίσω κάτι στο ελεκτικό συνέδριο. Καλό είναι να μας απαντάτε σε ερωτήσεις που δεν κάναμε, αλλά εγώ κάτι άλλο ρώτησα. Κάνετε μια ειδική έκθεση για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση και σε αυτή την ειδική έκθεση προσπάθησα να σα ζητήσω κάποια πράγματα να γράψετε εκεί. Επιθυμίε εξέφρασα, ε, σα παροτρύνω, πούμε, το κόστο τη πρόληψη προσωπικού της πρόσληψης ε, των ειδικών εκπροσώπων. Δεν ξέρω αν τα κατάλαβε το ελεκτικό συνέδριο. Αυτό θέλω να μου απαντήσετε. Δηλαδή τόσο περίεργα τα είπα και συγκεκριμένα και δεν τα καταλάβατε, γι' αυτό το επαναλαμβάνω τώρα. Ωραία. Θα Αφήσουμε το ελεκτικό συνέδριο να το σκεφτεί και να απαντήσει πρώτα ο κύριος Σάλιβαν στις άλλες ερωτήσεις του κυρίου Σικέρσκη και του κυρίου ε, Οντί. Ε, uh, uh, ναι κύριε Σικέρσκη, η σύντομη απάντηση είναι ναι, έχουμε απεσπασμένους εμπειρογνώμονες ή ειδικού από τις Γενικές Διευθύνσεις της Κομισιόν στις διάφορες αντιπροσωπείες μας, όχι όσους θα θέλαμε. Αυτό αποτελεί τεράστια πρόκληση, διότι αντιμετωπίζει δυσκολίε τελέχουση η Κομισιόν αυτή τη στιγμή. Θα θέλαμε φυσικά πάντα να έχουμε περισσότερου ειδικού από ε, γενικέ διευθύνσει όπω την ενέργεια ή την ε, έρευνα ή τι εσωτερικέ υποθέσει ή τη δικαιοσύνη. Η Κομισιόν κάνει κάποιες επιπλέον προσπάθειες για να διαθέσει κάποιες ε, επιπλέον θέσεις φέτος ώστε να αντιμετωπίσουμε την, ε, ε, το φόρτο εργασία που έχει αξιολογηθεί ότι θα υπάρξει με κάποια επανακατανομή προσωπικού της Κομισιόν. Η Κομισιόν δεν μπορεί να διαθέσει όσους θα θέλαμε. Αλλά τονίζω ότι συνεργαζόμαστε στενά και με τη Γενική Διευθυνσία Εσωτερικών Υποθέσεων στην αντιπροσωπεία μας στη Μόσχα. Έχουμε κάποιον υπεύθυνο για την ενέργεια, ο οποίος έχει στενή επαφή με τη Γενική Διευθύνση Ενέργειας της Βρυξέλλες, διότι φυσικά προωθούμε τις πολιτικές της Ένωσης μεταξύ των οποίων και αυτές για τις οποίες είναι υπεύθυνοι οι Επιτροπή στις δραστηριότητε μας. Αν μου επιτρέπετε κύριε Οντή, επίσημα το Κοινοβούλιο καλείται να χορηγήσει απαλλαγή για τις διοικητικές δαπάνες της ΕΙΕΔ για τις οποίες η κυρία Άστον είναι υπεύθυνη ως ύπατη εκπρόσωπος. Αυτό είναι ένα ξεχωριστό κεφάλαιο. Επίσης καλείστε να δώσετε και μια γνωμοδότηση για τον προεπολογισμό που έχω στην ε, Επιτροπή που αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα και για τον οποίο πάλι έχει αρμοδιότητα η κυρία Άστον ως αντιπρόεδρος. όπως και για το μέσο εξωτερική εξωτερικής πολιτικής. Μια υπηρεσία που δουλεύει υπό την κυρία στον έχουμε αυτή τη διαμόρφωση, διότι η συνθήκη δεν επέτρεψε, σύμφωνα με την Κομισιόν, τη μεταφορά της αρμοδιότητας για τη διαχείριση ορισμένων προπολογισμών απευθεία στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Επίσημα το αντικείμενο των συζήτησης μας σήμερα, αν έχω καταλάβει καλά, είναι ουσιαστικά οι διοικητικέ δαπάνε τη Υπηρεσία Εξωτερική Δράση. Φυσικά καταλαβαίνω ότι όλα αυτά πρέπει να ενταχθούν όπω είπε η κυρία Άστον. Δεν μπορούμε να αποχωρήσουμε, να ξεχωρίσουμε αυτό τον προπολογισμό από την εξωτερική δράση της Ένωσης που είναι ένα ζήτημα πιο ευρύ. Προσπαθήσαμε και μαζί και με το ελεγκτικό συνέδριο που εξέτασε τους λογαριασμούς να σας ε, διασφαλίσουμε, να σας διαβεβαιώσουμε ότι τα χρήματα που μας εμπιστευθήκατε για τις διοικητικέ δαπάνε τη υπηρεσία εξωτερική δράση ε, ε, ξοδεύτηκαν σωστά και χρησιμοποιήθηκαν σωστά. Αυτά μπορώ να σας πω εγώ εκ μέρους της ΕΕΔ. Φυσικά υπάρχει ένα πιο ευρύ πολιτικό περιβάλλον που εκτιμώ ιδιαίτερα, αλλά δεν εμπίπτει στι αρμοδιότητές μου. Ε, Ωραία. Ε, θα ήθελα να απαντήσει ο κύριο ε, Σίπινγκστον. Στα γερμανικά ο κύριος Πίνξτεν. Και βέβαια κυρία Γκρέσλε, σας καταλάβαμε πάρα πολύ καλά και εγώ και ο συνάδελφος Φαζάκας. Αλλά δεν πήραμε απόφαση για το τι θα βάλουμε στην ειδική έκθεση, ούτε το συγκεκριμένο πεδίο που θα καλύπτει ε, βεβαίως και σημειώσαμε τις ερωτήσεις, τουλάχιστον εγώ τις κατανόησα απολύτως. Όσο και ο κύριος Φαζάκας από ό,τι μου λέει. Πολύ ε, προσεκτικά σας ακούσαμε και σας ευχαριστούμε για τις ερωτήσεις σας. Ο Πρόεδρος. Ωραία. Ολοκληρώνεται εδώ αυτή η συζήτηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριο Σάλιβαν. Ε, λοιπόν, ακολουθούμε ε, τώρα το επόμενο θέμα. Περνούμε στην ψηφοφορία μας. Ε, είναι η γνωμοδότηση του κυρίου Ζαν για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ετήσια έκθεση 2011. Oui. Ορίστε κύριε Γκάιερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Από τη σκοπιά της δικής μας πολιτικής ομάδας μπορούμε να ψηφίσουμε όλα μαζί, αν μπλοκ, Όλες τις τροπολογίες του κυρίου Οντί, αλλά και όλες τις τροπολογίες της κυρίας Χέτζοκ. Δηλαδή σε ό,τι αφορά τους σοσιαλιστές και δημοκράτες μπορούμε να το διεκπαιρεώσουμε με μία και μοναδική ψηφοφορία. Ευχαριστώ πολύ λέει ο Πρόεδρος. Βλέπω εδώ ότι έχουμε προβλέψει στο κατάλογο ψηφοφορίες δύο ψηφοφορίες αν μπλοκ. Ε, συμφωνείτε να ψηφίσουμε έτσι. Ε, τις τροπολογίες πρώτα του εισηγητή 1 με 10 και μετά ε, τις τροπολογίες 11 μέχρι και 15 όπως βλέπετε στο δεύτερο μπλοκ. Σε δύο ενότητες λοιπόν, όχι μία ενιαία ψηφοφορία. Ψηφίζουμε το πρώτο μπλοκ 1 με 10. Ψήφι κατά, αποχές, εγκρίνονται. Περνάμε τώρα στη δεύτερη ενότητα, 11 με 15 ομού οι τροπολογίες, ψήφι κατά, αποχές, κανείς ε, αντίθετος, εγκρίνονται. Και ψηφίζουμε τώρα το σύνολο ηλεκτρονικά, το σύνολο του σχεδίου γνωμοδότησης όπως τροποποιήθηκε. Πέρασε. Μάλλον όχι, τώρα αρχίζει η ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι. Πέρασε. 14 ψήφοι υπέρ, καμία ψήφος κατά, καμία αποχή ομόφωνα. Συγχαρητήρια κύριε Ντί. Εγκρίνεται το σχέδιο γνωμοδότησής σας. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία. Α, ορίστε κύριε Ντί, έχετε το λόγο. Ναι, θα ήθελα μόνο να ευχαριστήσω τους συναδέλφους και τους σκιώδης εισηγητές, τη γραμματεία αλλά και τις υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων που με βοήθησαν ε, να αποφύγω κάποια ασφάλματα στην εκτίμησή μου και στη βελτίωση της νομοδότησης που θα διαβιβαστεί στην Οικονομική Επιτροπή. Και θυμίζω ότι εμείς έχουμε την αρμοδιότητα βάσει κανονισμού για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, κύριε Πρόεδρε. Να σας ευχαριστώ και εγώ, Ο Ζωμπιέρ. Λύεται η συνεδρίαση, η προσεχή συνεδρίαση είναι στι 21 Ιανουαρίου στις Βρυξέλλες στις 3 το μεσημέρι και στις 22 Ιανουαρίου και στις 24 όπως βλέπετε στη μέση διάταξη. Σας ευχαριστώ πολύ χαίρετε.